So, Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Ε, θα ψηφίσουμε σήμερα με, με ασυνήθιστο τρόπο ε, ε, στη στρογγυλία του τη αίθουσα, όπως συνήθως έχουμε τη, τους τριμερείς διαλόγους μας. θα πρέπει να το συζητήσουμε και με τους ε, συντονιστές μας, ε, διότι δεν μπορεί η μεγαλύτερη νομοθετική επιτροπή του Κοινοβουλίου ε, να πρέπει λόγω κάποιας ακρόασης ε, να εξωθείται από την αίθουσα. Θα πρέπει να μιλήσουμε με τη διοίκηση, να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι που μας έχουν βάλει εδώ πέρα. Προχωράμε λοιπόν. Με το ψήφισμα για το site COP16 ξεκινάμε με την τροπολογία 1 και έχουμε την παράγραφο 9. Ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ σκώστε τα χέρια σας. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22, χωριστή ψηφοφορία, πρώτο μέρος, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε στο δεύτερο μέρος της τροπολογίας 22. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές Δεν μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, να το ελέγξουμε αυτό ηλεκτρονικά. Το δεύτερο μέρος στις 22. Haben Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 16 κατά. Το δεύτερο μέρος της 22 εγκρίνεται. 24 υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές, ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 25, αρχή της ψηφοφορίας. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 18 κατά εγκρίνεται, 26 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται, 27 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται, 28 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται, 29 Ε, ε, καταπίπτει η 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 31 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, 32 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, μόνο οι σοσιαλδημοκράτες υπερψηφίζουν, οι άλλοι απεργούν. Oral amendment to amendment 37. Ε, τροπολογία 37. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να το ελέγξουμε. Ψήφισαν όλοι. 27 ε, υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται. Ε, η 37 υπέρ, κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει η 23 και φτάνουμε στην 40 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 43 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46. Δεν είναι απαραίτητο να την ψηφίσουμε. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 Κατά πίπτη 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ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 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Την 10, ηλεκτρονικό έλεγχο. ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 30 υπέρ 22 κατά εγκρίνεται. 13. Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεκατέσσερα. Υπέρ. Κατά. Το δεύτερο μέρος καταπίπτει, λέει ο πρόεδρος, στις 13. Γι' αυτό ψηφίζουμε την 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18. Καταπίπτει 16. Ελέγχουμε τη 15 μάλλον. 15. 15. Τη 15 ελέγχουμε. Ψήφισαν όλοι. Λήξη τη ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 23 κατά. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 56 υπέρ, κανείς κατά, καμία αποχή, θερμά συγχαρητήρια στους συντάκτες αυτού του ψηφίσματος.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 Θα ξεκινήσουμε με τη νομική βάση που τροποποιείται με την τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε στην τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 14. Υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε τη 14 ηλεκτρονικά αρχή της ψηφοφορίας 14 ψήφισαν όλοι λήξη της ψηφοφορίας 33 υπέρ 27 κατά εγκρίνεται Ψηφίζουμε την τροπολογία 54 με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ? κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Dann consolidated amendment 5. Wer ist dafür? Ενοποιημένη τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 13 καταπίπτει, 18 και 14 είναι όμοιες, ε, ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 67. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 36 κατά, απορρίπτεται. Ενοποιημένη 6 υπέρ. Ενοποιημένη 7 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 8 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπέρ. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 20 καταπίπτει. Ήτρε 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την Ήτρα 18 ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 40 κατά, απορρίπτεται σαφώς. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ποιος ζήτησε έλεγχο? Ακόμα ε, ε ψηφίζαμε, δεν μπορούμε να ελέγχουμε ταυτόχρονα. Ήτρα 19, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 75, υπέρ. 75, υπέρ. Κατά. Ε, υπέρ μάλλον, κατά. Απορρίπτεται. 21 η εκρίνεται απαράδεκτη. Φτάνουμε στην ενοποιημένη 9. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 22 υπέρ. 22 καταπίπτει. και η 83 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρο της 32 έχει αποσυρθεί. 85 και 32 μέρο 3 τις ψηφίζουμε μαζί. Ποιες είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 το τέταρτο μέρο έχει αποσυρθεί. 86 καταπίπτει. Και η άλλη καταπίπτει. 88 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Ε, αποχές δεν είναι σαφές. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 34 υπέρ, 29 κατά. Ε, ψηφίζουμε την 34. Ε, Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 37-38 έχουν αποσυρθεί. 89 και 90 τις ψηφίζουμε μαζί. Ποιες είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 39 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε στα εκτιμώντα, τροπολογία 3 υπέρ. Κάποιο ε, θέλει να ελέγξουμε την 39, ελέγχουμε ηλεκτρονικά αρχή ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι.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 κατά από αποχές εγκρίνεται. Η 7 έχει αποσυρθεί, 48 υπέρ κατά από αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 2 υπέρ κατά από αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 53. Αρχή της ψηφοφορίας. Haben alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται 32 υπέρ 28 κατά. Dann geht's weiter mit 7, ITRE 7. ITRE 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία πάνω στην πρόταση όπως έχει τροποποιηθεί. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας 64 υπέρ, και τελική ψηφοφορία πάνω στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος στο σύνολό του. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Μία ψήφος κατά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θερμά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Dann kommen wir jetzt zum This was a tricky thing. Yeah, let's, Ist nicht zulässig, ne? Let's see if anybody says anything. Wir stimmen dann ab über den Bericht Rossi. Ψηφίζουμε τώρα την έκθεση Ρώση. Δεν ψηφίζουμε την 1, διότι κρίθηκε απαράδεκτη. Ψηφίζουμε την 5. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 Ρόσπαχ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συνάδελφος Ρότε Μπέρεντ ε, ε, μίλησε λιγότερο από τον συνάδελφο Σνέλχαρτ σήμερα το πρωί. Κάτι της χρωστάω Πέτη 5-2 υπέρ. Κατά. Αποχές Πέτη 5-3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 46. Αρχή της ψηφοφορίας ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 32 υπέρ, 29 κατά, 47 ε, υπέρ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 Κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 58, 59 και 60 και φτάνουμε στην 61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πέτει 6, β υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές, το ελέγχουμε. 65. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας.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 όχι, πρέπει να την ψηφίσουμε. 78 ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. απόχε εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. 112 καταπίπτει. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82-83 τις ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνονται. 84 καταπίπτει. Πέτη 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 98 Ψήφισαν όλοι η λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 100. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 34 υπέρ 29 κατά. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 112 έχει αποσυρθεί. 113 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ δεν, δεν εγκρίνεται. Ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 5η 5. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 39 κατά. Έχει δίκιο. 5-8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 8. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 8. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Ο Χωσνέλχαρτ δεν έχει δίκιο, εγκρίνεται. Εγκρίθηκε. Πέτει 9, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται. 23 καταπίπτει. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά Δεν ήταν σαφές. Παρακαλώ να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 41. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται σαφώς. Η ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 63 υπέρ. Ο Κάνχαϊντς Φλόρεν ζητάει το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση έχει τώρα διαφορετικό πρόσωπο και γι' αυτό δεν ε, την καλύπτει πια η αιτιολογική έκθεση που έγραψε αρχικά ε, ο εισηγητής. Ε, παρακαλώ λοιπόν την Επιτροπή να, μου, να δεχτεί να γράψω εγώ μια αιτιολογική έκθεση που να αντιστοιχεί σε αυτά που ψηφίσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση αυτή ότι ο εισηγητής ε, θα πρέπει να προσαρμόσει το μέρος αυτό. Εάν δεν το κάνει ο εισηγητής θα διαγραφεί τελείως. Εντάξει, ωραία. Προχωράμε. Wir kommen jetzt zum Bericht und Φτάνουμε στην έκθεση Λιωτάρ. Και ξεκινάμε με την ενοποιημένη τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πηδάμε στην τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε στην ενοποιημένη 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3β ε, νέο, τροπολογία 35, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 36, χωριστή ψηφοφορία, το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, απόχε εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 το δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. 38 το δεύτερο μέρος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40. Προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Ενοποιημένη 4 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Ενοποιημένη 5 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 51 το πρώτο μέρο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ενοποιημένη 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 57 με προφορική τροπολογία σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, ένα μέρος έχει μόνο. 6β νέο τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ενοποιημένη 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 15, ενοποιημένη 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 118 το πρώτο μέρο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 118 το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 108. Χωριστή ψηφοφορία σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. 110 ψηφίσουμε ηλεκτρονικά αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έμπλη 15 υπέρ. Να ελέγξουμε την 129 αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε, λήξη της ψηφοφορία. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν μία ψήφο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Λήξη της ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 26 κατά, 5 αποχές. Εγκρίνεται. Φτάνουμε στην έμπλη 15. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 16. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 133. Υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εμπλεπτά υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει η 131 και φτάνουμε στην έμπλη 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 με προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 έμπλη Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, φτάνουμε στα εκτιμώντα. τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2. Τις ψηφίζουμε μαζί, 2 και 3, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 4 και 5 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 6, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 7, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική όπως πάντα, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι, λήξη της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας. 62 υπέρ, μία αποχή. Θερμά συγχαρητήρια στην κυρία Λιωτάρτ. Thank you very much. And now we have endocrine disruptors. So you're okay. Dann kommen wir zum Initiativbericht von Orsa West φτάνουμε στην, ε, στην ε, έκθεση πρωτοβουλίας ε, της κυρίας Βέσλουντ και ξεκινάμε με την τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένοι 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 48 πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ενοποιημένη 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 70. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ενοποιημένη 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κατά πίπτη 86, φτάνουμε στην 87, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 88, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται, αλλά να ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι η λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 110. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία, 34 υπέρ, 27 κατά. 111 υπέρ, κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές αυτό, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ, λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ενοποιημένη 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 138 σε δύο μέρη, το πρώτο μέρος, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 139. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 δεν πρέπει, χρειάζεται να την ψηφίσουμε και φτάνουμε στην 156 το δεύτερο μέρος ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία είναι αποσύρθηκε Φτάνουμε στην τροπολογία 2. Όχι, λάθος. Τροπολογία 3, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έτσι δεν είναι. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 3, για να είμαστε σίγουροι. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται σαφώς. Ε, πότε, πότε κάποιοι, κάποιος σου παίρνει ο ύπνος, γι' αυτό διακόπτουμε λίγο. Ε, τροπολογία 4, υπέρ. Κατά. Τρεις ε, συνάδελφοι συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Ε, ελέγχουμε. Τροπολογία 4, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, εγκρίνεται, διορθώνει ο Πρόεδρος. Και, και εγώ μου φαίνεται κοιμάμαι, λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 6, υπέρ. Κατά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 Ενοποιημένη 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ελέγχουμε την 21 ηλεκτρονικά αρχή της ψηφοφορίας ψήφισαν όλοι παρακαλώ λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται φτάνουμε στην 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να το ελέγξουμε Ελέγχουμε την 27 ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχή ψηφοφορία. ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι η λήξη της ψηφοφορίας. 55 υπέρ, 6 κατά, μία αποχή. Θερμά συγχαρητήρια στην Όσα Βέσλοντ. Wir kommen jetzt zur Entlastung. Φτάνουμε στις απαλλαγές για τους διάφορους οργανισμούς. Η συγγήτρια είναι η Γιούτα Χάουκ. Ε, τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας.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 Απαλλαγή για το τμήμα 3 του προπολογισμού και πάλι είναι η συγκήτρια η Ιούτα Χάουκ. Τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Ε, ζητούν έλεγχο για την τροπολογία 1. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 6 υπέρ. 55 κατά. Απορρίπτεται σαφώς. Τροπολογία 2. Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελεκτική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. «52 υπέρ Αυτά κατά εγκρίνεται». Ευχαριστούμε πολύ την Γιούτα Χάουκ. Και πάλι Γιούτα Χάουκ. Αυτή τη φορά ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Ε, τροπολογία 1. ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Συγγνώμη, για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη και Ελέγχου Νόσων. Ε, τροπολογία 2 με προφορική τροπολογία. ποιο είναι υπέρ. Ποιο είναι κατά. αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη τη ψηφοφορία 55 υπέρ, 5 κατά, καμία αποχή. Ευχαριστούμε πολύ Γιούτα Χάουκ. Wir Φτάνουμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, λέει ο πρόεδρο. Ε, πάλι Γιούτα Χάουκ. Έχουμε τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται.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 Αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξτε της ψηφοφορίας. 53 υπέρ. 4 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται σαφώς λοιπόν. Damit kommen wir zur Umweltagentur, zur Haushaltsentlastung und zwar ab. Απαλλαγή για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται με προφορική τροπολογία. 5, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 8 ψήφους κατά και 54 υπέρ. Φτάνουμε στην ΕΦΣΑ, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ένα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρία. Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Πέντε υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6. Με προφορική τροπολογία της εισηγήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 ε, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 13 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική οριστική, ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνεται 46 υπέρ, 14 κατά. ΕΜΑ, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Με προφορική τροπολογία τη συγγήτρια, ε, Ποιο είναι υπέρ, κατά, Αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ. Κατά. απόχέ απορρίπτεται. Τροπολογία 4 σε δύο μέρη, πρώτο μέρο υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική, οριστική, ε, τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. 52 υπέρ, 8 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. So, Kollegen und Kollegen, vielen, hm? vielen Dank. Es geht jetzt weiter im Text und zwar mit. Ε, προχωράμε στο σημείο 19. Την έκθεση του Κάρλ Σλίτερ. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Παρακαλώ. When is the minister coming? Five. Five o'clock. Five. Five. Yes. Is the minister coming at five? So, alle, die an der Aussprache teilnehmen möchten, teilnehmen möchten. Παρακαλώ όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στην συζήτηση για την ανακύκλωση των πλοίων είναι ευπρόσδεκτοι όποιοι θέλουν ε, να ασχοληθούν με άλλες δραστηριότητες ε, μπορούν ε, στις 5 η ώρα περιμένουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος της Ιρλανδίας. Θα εξετάσουμε λοιπόν πρώτα την έκθεση του Καρλ Σλίτερ. Έχεις το λόγο, Καρλ. Yeah. Well, you don't need to leave, all of you. It's really interesting dossier. It's the... Μην φεύγετε όλοι, είναι πολύ ενδιαφέρον ε, το θέμα για την ανακύκλωση των ε, σκαφών. Ε, Βεβαίω στην Ευρώπη το 90% των κατόχων πλοίων δεν ενδιαφέρονται καν για την νομοθεσία. Εμείς ουσιαστικά θέλουμε να πείσουμε τους πολίτες να εφαρμόσουν αυτή την νομοθεσία γιατί είναι πολύ καλή νομοθεσία που θέλουμε να εφαρμοστεί. Παρακαλώ, ε, ησυχία να επικρατήσει την αίθουσα και όσοι δεν θέλουν να παραμείνουν να αποχωρήσουν. Excuse me. Okay, Mr. Schlitter, it's, the floor is yours again. I heard Rod complaining it's not exciting enough. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ δελεαστικό το θέμα, τουλάχιστον έτσι νομίζετε. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και συναρπαστικό ζήτημα. Ποια, πώς έχει κατάσταση σήμερα Ακριβώς επειδή δεν ε, επεξεργαζόμαστε ε, τα απόβλητα όπως ε, πρέπει, έχουμε τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις με τεράστια εξωτερική ανάθεση του κόστους μόνο και μόνο για εξοικονόμηση μερικών μικρών χρηματικών ποσών. Εδώ και 14-15 χρόνια υπάρχει απαγόρευση αυτής της πρακτικής έτσι κι αλλιώς τα σκάφη έχουν, πάντα περιέχουν ε, επαρκή επίπεδα ε, βλαβερών αποβλήτων. Παρ' όλα αυτά δεν λειτουργούν οι κανόνες αυτοί. Η κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ άσχημη. Η πλειονότητα των ε, πολιτικών ομάδων ε, επιθυμεί να βρει ένα καλό τρόπο ε, να λειτουργεί πολύ καλύτερα η ανακύκλωση των σκοφών. Οι περισσότερες ομάδες έχουν καταθέσει τροπολογίες με στόχο να υπάρχει ένα είδος χρηματοδοτικού μηχανισμού για να επιβάλλεται αυτή η νομοθεσία. Έχει γίνει και η πρώτη συνεδρίαση των σκιωδών και δεν ήταν εύκολο να βρούμε τον έναν και μοναδικό μηχανισμό με τον οποίο θα συμφωνούν όλοι. Όμω, μπορούμε να πούμε ότι η πρόταση της Επιτροπής ε, δεν ε, τη χάνει τη στήριξη ε, της πλειονότητας των ομάδων, ε, θεωρούν ότι δεν είναι επαρκής και υπήρξε και μια ένταση για να αποφευχθεί το outflagging, δηλαδή η εγκατάλειψη των κοινωτικών νεολογίων και υπάρχουν και κάποια νομικά ζητήματα. Γι' αυτό ζητήσαμε από την νομική υπηρεσία να απαντήσει κάποια από αυτά τα ερωτήματα. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν αν αυτό που κάνουμε θεωρείται νόμιμο εφόσον έχουμε αυτή την απαγόρευση εξαγωγής, είναι νόμιμο να έχουμε εξαίρεση. Η νομική υπηρεσία έκανε μια γνωμοδότηση. Βέβαια, ίσως είναι εμπιστευτική, δεν ξέρω αν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά μπορούμε να τους ζητήσουμε να μας πούν αν θέλουν. Το βασικό συμπέρασμα είναι όμως ότι αυτό που κάνουμε είναι νόμιμο. Ιδίως καθώς ο σκοπός ε, της απαγόρευσης της βασαλίας ήταν ε, να μην υπάρχει αυτή η μη ικανοποιητική διαχείριση ε, στις τρίτες χώρες. Και αν αυτή η επεξεργασία είναι εντάξει, είναι σωστή, τότε είμαστε κι εμείς εντάξει με τα κριτήρια μας. Όμως θα ήταν χρήσιμο και για την νομική υπηρεσία να μας διαφωτίσει λίγο για την τροπολογία που είχε κατατεθεί να διαγραφεί από το άρθρο 29. Ποιες θα ήταν λοιπόν οι νομικές επιπτώσεις της διαγραφής αυτής της ε, συγκεκριμένης ε, εξαίρεσης και της τροποποιημένης ε, εξαίρεσης που πρότεινα εγώ εφόσον θεωρούμε ότι πριν φύγει και όλες από τα ίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται απόβλητα. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε να δώσουμε το λόγο στην νομική υπηρεσία ποιος, ε, ποια είναι η νομική συνέπεια της διαγραφής της εξαίρεσης από το άρθρο 29. Στη συνέχεια, το άλλο ζήτημα είναι, ακόμα και αν όλοι συμφωνούμε επί του χρηματοδοτικού μηχανισμού, τι συμβαίνει ε, με τις δικές μας ε, αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν έχουμε τέτοιο μηχανισμό. Αυτός ο μηχανισμός δηλαδή ε, θα δίδει κονδύλια μόνο αν υπάρχει η διάλυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον ΩΣΑ ή θα έχουμε έναν κατάλογο με εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο. Το πώς θα εξετάσουμε αυτό το ερώτημα μας επηρεάζει για το τι θα γίνει με το Ταμείο ή αν υπάρχει ένα, ε, ένας μηχανισμός ασφάλισης ή και τα δύο. Γιατί αν ζητάμε από όλους να πληρώνουν και δίδουμε χρήματα μόνο αν γίνεται η διάλυση από συναρμολόγηση στην Ευρώπη, τότε υπάρχουν επιπτώσεις. Όμως αν βρούμε νόμιμο τρόπο να γίνει αυτό, για παράδειγμα μόνο ε, τα ευρωπαϊκά σκάφη να πληρώνουν, τότε υπάρχει ο κίνδυνος του, της εγκατάλειψη των κοινωτικών νεολογίων outflagging. Αν όμω βρούμε τρόπο να, να γίνεται αυτό νόμιμο και να τα δίνουμε και πάλι στην Ευρώπη, ο χρηματοδοτικό μηχανισμός θα είναι πολύ πιο ακριβώ. γιατί η διαφορά κόστους που θα, πρέπει να καλυφθεί, όλο το νόημα τέτοιων ε, μηχανισμών είναι να μην δίνουμε κίνητρο σε κάποιον να παρανομεί. Να είναι ε, ε, προς το συμφέρον του άλλου να εφαρμόσει τον νόμο. Άλλη επιλογή είναι να μη συμμετέχουν όλες οι χώρες, αλλά όσο χώρες του ΩΣΑ. Τότε η διαφορά θα είναι μικρότερη ή να έχουμε κάποια πρότυπα. Όμως αυτό μετά επηρεάζει και τις θέσεις εργασίας που κάποιοι θέλουν από τους σκιώδεις. Πρέπει να βρούμε λοιπόν ε, μια καλή ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία. Άλλη εναλλακτική είναι να καλυφθεί η διαφορά κόστους από την αξία του μετάλλου που ε, παίρνουμε ουσιαστικά μετά τη διάλυση του πλοίου. Αλλά και αυτό μετά έχει σχέση με τον έλεγχο και την καταβολή πόρων από το Ταμείο. Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές τιμών ε, ένα σκάφος πάντα έχει κάποια αξία στο τέλος της ζωής του γιατί έχει ήδη πολλά υλικά μέσα και μέταλλα. Όμως η τιμή είναι πολύ διαφορετική αν έχουμε ε, χαμηλά αμοιβόμενου εργαζομένους με κακές, ε, κακούς όρους εργασίας. Έχουμε λοιπόν πολλέ πρακτικέ όπω η προσάραξη. Αν θέλουμε κατάλληλε εγκαταστάσει με καλά αμοιβόμενου εργάτε, ε, θα πρέπει κάποιο να καταβάλει πολύ μεγαλύτερο ε, ποσό για την αποσυναρμολόγηση. Είναι πολύ σημαντική η διαφορά. Ακόμα και τα 200 ευρώ ανατόνο φτάνει αυτή η διαφορά λοιπόν. Ε, ανάμεσα σε τι θα πληρώσει κάποιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποσυναρμολόγηση και σε μια προσάραξη στο Μπαγκλαντέ. Όμω, αν έχουμε αυτό το συνολικό σχήμα, το μηχανισμό, ίσως ακόμα και το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές ε, να πληρούν ε, τα κριτήρια με συγκεκριμένους ε, μηχανισμούς που και πάλι θα είναι ε, αποδοτικοί. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιε εγκαταστάσει ακριβώ θα μπουν στον κατάλογο. Κατά τη γνώμη μου, ο Ευρωπαϊκό Κατάλογο θα αναφέρει ποιε εγκαταστάσει πληρούν τα κριτήρια ε, για ένα σοβαρό και ασφαλέ ε, περιβάλλον αποσυναρμολόγηση με παράλληλη προστασία των εργαζομένων. Οποιαδήποτε χώρα ε, μπορεί να τηρεί αυτές τις προδιαγραφές, για μένα πρέπει να μπαίνει στον κατάλογο. Και έτσι αποφεύγουμε τις κακές πρακτικές ε, με κακά αμοιβόμενου εργαζόμενου, αλλά και για τις επιπτώσεις για τη φύση. Έχουμε μακρά παράδοση με όλη αυτή την ιστορία και στη χώρα μου και αλλού. Ε, και στη χώρα μου πλέον δεν είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό. Ρίξαμε εκατομμύρια ε, σε αυτή τη βιομηχανία και παρόλα αυτά σήμερα 1,5% της ε, χωρητικότητας, της παγκόσμιας χωρητικότητας, 2,5 μάλλον, διορθώνω, ε, κατασκευάζεται στην ε, Ευρώπη. Γιατί έχουμε ακόμα σημαντικό μερίδιο της αγοράς ε, στα σκάφη πολυτελείας. Ενώ 95% είναι στην Κίνα, στην Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ακόμα ικανότητες από στην Ευρώπη και είμαι διατεθειμένος να εξετάσω πώς μπορούμε να διατηρήσουμε αυτές τις εγκαταστάσεις που να μην κοστίζουν βέβαια ε, δυσθεώρητα ποσά και να είναι και νόμιμες βέβαια αυτές οι εγκαταστάσεις. Βασική όμως προτεραιότητα είναι αυτές οι εγκαταστάσεις να είναι ασφαλείς. για τα σκάφη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η βασική η αρχική μου πρόταση ήταν να υπάρχει ένα ταμείο το πλεονέκτημα αυτού του ταμείου είναι ότι μειώνει τον κίνδυνο απάτης, ε, outflagging, ανακατάληψη ε, των κοινοτικών νεολογίων, δεν επιφέρει επιπλέον διοικητικό άχθος και είναι εύκολα εφαρμόσιμο και άμεσα εφαρμόσιμο. Όμως, το μειονέκτημα είναι ότι δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στα υπόλοιπα σκάφη εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν το ότι δεν υπάρχει ε, κίνητρο για το outflagging. Ε, γι' αυτό ο Chris Ντέιβι και οι φιλελεύθεροι ε, πρότειναν ένα συνδυασμό των δύο που θα έχουμε κάποιο είδους ασφάλιση για να γίνεται καλύτερη διάλυση των σκαφών και έτσι θα μπορούμε αυτό να το πειράσουμε. Ωστόσο, είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τα, κριτήρια που θα βάλουμε στις χώρες ε, μη, ε, που είναι εκτός του ΩΣΑ πέραν των προδιαγραφών ε, της συνθήκης της Βασιλείας. Επιμένω επίσης ότι οποιοδήποτε μηχανισμός δεν πρέπει να δίνει κριτήρι, κίνητρο συγγνώμη, για το outflagging. Εγώ λοιπόν προτείνω να βασίσουμε το συμβιβασμό μας στην εξή επιλογή. Να υπάρχει ένα ταμείο που θα είναι υποχρεωτικό για τα ευρωπαϊκά σκάφη να ε, πληρώνουν και σκέφτομαι και το εξή. Είναι δύσκολο για ένα σκάφος τρίτης χώρας που φτάνει, έρχεται μία φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει υποχρέωση για πλήρες ε, σχήμα ασφάλισης θα υπάρχει πρόβλημα να εφαρμοστεί αυτό διεθνώ. Γι' αυτό σκεφτόμουν να δοθεί η δυνατότητα στα σκάφη ε, τρίτων χωρών σημαία, όταν έρχονται στην Ευρώπη, είτε να δίνουν μια απόδειξη ε, οικονομικής ε, ασφάλισης, επειδή έρχονται συχνά, για παράδειγμα, ή επειδή έχουν άλλους ε, λόγους εμπορίας, ή να πληρώσουν το αντίτιμο όταν έρχονται, προσεγγίζουν το λιμένα. Και αυτό από νομική πλευρά τουλάχιστον δίνει τη δυνατότητα αυτή στα σκάφη τρίτη χώρα και πάλι δεν δίνουμε κίνητρο για το outflanking. Κάτι τέτοιο τέλο πάντων. Και μετά, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει πολύ πρόσφατα ε, μου παρουσίασαν μία πολύ καλή ε, μελέτη για τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού του ταμείου και γιατί πρέπει να πάμε προς ε, την άλλη επιλογή ε, της ασφάλισης. Θα εξετάσουμε τις προτάσεις τους και θα δούμε μήπως μπορεί να τροποποιηθεί καταλήλως και η τρέχουσα πρόταση. Επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί στην αρχική πρόταση έχουμε αυτή την, το insurance, αυτή την ασφάλιση, όμως αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, εν προκειμένου, γιατί Όπω αναφέρθηκε σήμερα από τι τροπολογίε, τροπολογίες, αναφορά στην οδηγία 2009-20 για την ευθύνη της ασφάλισης, insurance liability, εκεί μιλάμε για ασφάλιση απέναντι σε κάτι που δεν θέλουμε να συμβεί και γι' αυτό αναλαμβάνεται η ευθύνη ή πληρώνεται ένα αντίτιμο. Ενώ εδώ η ασφάλιση είναι για κάτι που θέλουμε να συμβεί. Είναι διαφορετική λογική λοιπόν. Ε, κατά πόσο είναι λογικό δηλαδή να ε, παραπέμψουμε στην ε, εν λόγω οδηγία 2009-20 ή μήπως πρέπει το χρηματοδοτικό μέσο 2020 ή μήπως πρέπει το χρηματοδοτικό μέσο να πάρει μια διαφορετική ονομασία. Αλλά καλό θα ήταν η Επιτροπή να μας απαντήσει σε αυτό. Εδώ θέλω να δώσω το λόγο στους ασκιώδεις εισηγητές και θα προσπαθήσω να αρχίσω τη σύνταξη των ε, συμβιβαστικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης ε, μιας ε, οικονομικής ε, ασφάλειας ή κάποιου χρηματοδοτικού μέσου. Εγώ κλείνω προς την πρόταση τη συνδυαστική για τις χώρες, για τα σκάφη τρίτων χωρών και διατήρηση του Ταμείου για τα Ευρωπαϊκά. Πρέπει να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση, γιατί προβληματισμός μου είναι μήπως δώσουμε τη δυνατότητα, μήπως ανοίξουμε την πόρτα στην απάτη ή τι είδους ε, ασφάλειες θα έχουμε για τους νέους ιδιοκτήτες. Μετά πρέπει να συμφωνήσουμε. Ξέρω ότι υπάρχει σημαντικό συμφέρον ε, να έχουμε κοινό μηχανισμό, αλλά να μην αποτελέσει και μειονέκτημα και ξέρω ότι αυτή είναι ανησυχία πολλών. Θα ακούσω λοιπόν τη συζήτηση. Ε, συναντήθηκα και με εκπροσώπους της ε, Προεδρίας. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ η προσέγγιση τους. Θα προσπαθήσουν και εκείνοι να ε, εξετάσουν το ζήτημα το συντομότερο δυνατόν, γιατί και εκείνοι θέλουν να βρεθεί μια καλή λύση για το πρόβλημα. Να αξιοποιήσουμε και εμείς λοιπόν την ευκαιρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Θα δώσω το λόγο τώρα στην νομική υπηρεσία. Ο κύριος Λούκα Βθάτσιο είναι μαζί μας, οπότε παρακαλώ και το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν συντομία να απαντήσω στο ερώτημα του εισηγητή. Η ερώτηση είναι ποιες νομικές συνέπειες πιθανής διαγραφής του άρθρου 29 της πρότασης κανονισμού. Το άρθρο 29 περιέχει τη διάταξη εκείνα που περιλαμβάνει τα πλοία, μάλλον αποκλεί τα πλοία ε, του κανονισμού από το σύστημα ε, Hong Kong. Είναι δηλαδή εναλλακτική. Ποιο σύστημα τα δύο θέλουμε. Περίπλοκο το ζήτημα. Πρώτη όψεω, να πω δύο βασικέ συνέπειε. Πρώτα απ' όλα για λόγου ασφάλεια δικαίου. Έχουμε δύο δέσμες κανόνων που εφαρμόζονται για τα πλοία που είναι προς παροπλισμό από την υπηρετήση ο κανονισμός μας και πρέπει να αφορά όλα τα επικίνδυνα απόβλητα δηλαδή και από την άλλη ο κανονισμός για τα πλοία που είναι συγκεκριμένα για τα πλοία και μόνο. Όταν ε, δεν υπάρχει ε, σύγκρουση δικαίου, δηλαδή δεν υπάρχει ειδική διάταξη που να μιλάει για ποιο σύστημα πρέπει να εφαρμόσει τον εργαστικά, τότε Πρέπει να είναι σαφές πότε το ένα εργαλείο υπερέχει του άλλου ή μπορούν να εφαρμοστούν ταυτόχρονα. Αυτό το ερώτημα παραμένει ανοιχτό, είναι καθαρά νομικό ερώτημα και πρέπει με κάποιον τρόπο να το απαντήσουμε. Η δεύτερη συνέπεια κατ' εμέ αφορά την, τον όλο στόχο της άσκησης Hong Kong. Κατά τη γνώμη μου, η σύμβαση του Χονγκ Κόνγκ και η πρόταση κανονισμού που θέλει ουσιαστικά να εφαρμόσει τη σύμβαση έχει σκοπό λοιπόν να δημιουργήσει ένα δικό καθεστώ για τα πλοία και να λειτουργεί εναλλακτικά σε σχέση με το, με το σύστημα της βασιλείας. Ακριβώ λοιπόν, πρέπει να δούμε ποιε είναι οι συνέπειε αυτού του ελεκτικού συστήματο. Ξέρουμε ότι το σύστημα τη Βασιλεία έχει συγκεκριμένε διατάξει περί παρακολούθηση, ελέγχου κτλ. Τη ίδιε Βασιλεία, τα συμβαλόμενα μέρη κάλεσαν τον IMO να προβεί σε συγκεκριμένου κανονισμού για την ανακύκλωση των πλοίων. Και πάμπολε φορέ έχουν πει ότι δεν πρέπει να υπάρχει επικάλυψη κανονισμών για το ίδιο θέμα. Αυτό το τι δείχνει ότι τα δύο συστήματα λειτουργούν ή πρέπει να λειτουργούν εναλλακτικά. Οπότε λέω εγώ, ακόμα και αν η ταυτόχρονη εφαρμογή των δύο ε, συμβάσεων Hong Kong και πρόταση κανονισμού προκειμένου, νομικά καθαρά και μόνο, η ταυτόχρονη εφαρμογή τους εννοώ, θα μας επιστρέψει στο status quo. Τα προβλήματα δηλαδή που αντιμετωπίζονται αυτή τη στιγμή σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος βασιλείας θα συνεχίσουν να υπάρχουν και ο όλος στόχος αυτής της άσκησης που ήταν για η αναδιατύπωση της Χογκόν και να προτείνουν την, ένα κανονισμό για την ακύκλωση των πλοίων ουσιαστικά θα έχει ιτηθεί. Γιατί θα παραμένει το ίδιο πρόβλημα. Αυτά έχω να πω προκαταρτικά. Ευχαριστώ. Vielen Dank und dann steigen wir ein in Ευχαριστώ πολύ. Και θα ακούσουμε τώρα του σκιώδει εισηγητέ. Ο Κρίστοφερ Φιέλνερ ζήτησε πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ένα πρόβλημα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Έχουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά τη διάλυση των πλοίων και ε, ως απάντηση ε, παγκόσμια σε αυτό ε, είχαμε τη σύμβαση του Χονγκ Κονγκ. Ε, γι' αυτό έχουμε και το θέμα της πρότασης της Κομισιόν αλλά ο κύριος Σλίτερ και άλλοι συνάδελφοι ε, ισχυρίζονται ότι η σύμβαση του Χονγκ Κονγκ δεν αρκεί διότι έχει πολλά παραθυράκια. Είναι σαν ε, ελβετικό τύρι, πιο πολλές τρύπες. Έχει παρατηρεί. Η πρόκληση που βλέπω εγώ εδώ είναι ότι μάλλον είναι σωστό αυτό. Μπορεί να μην αρκεί η σύμβαση του Χονγκ Κόνγκ. Είναι δύσκολο να το δούμε αυτό ε, προτού να την εφαρμόσουμε. Μάλλον δεν αρκεί όμως, μάλλον θα χρειαστεί κάτι παραπάνω. Και έτσι έχουμε δύο επιλογές. Ε, είτε θα δημιουργήσουμε ένα ταμείο, είτε θα επιτέξουμε ένα μοντέλο ασφάλισης. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να επιλέξει κανείς ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Ε, ανάμεσα σε αυτές τις προτάσεις που ακούω από τους συναδέλφους, διότι ειλικρινά, δεδομένου του χρόνου που είχαμε να μάθουμε, να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες, να έχουμε ακροάσεις κλπ, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέρμα. Ε, και μιλάμε για επιλογή ανάμεσα σε δύο αρκετά διαφορετικούς δρόμους. Αφού όμως αποφασίσουμε αν θα επιλέξουμε ταμείο ή πρόγραμμα ε, ασφαλιστικό, θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιο πληρώνει, ποια ε, πλοία είναι υποχρεωμένα να συνεισφέρουν ε, και θα πρέπει να συνεισφέρουν μόνο αυτά με ευρωπαϊκή σημαία ή όλα. Και όπως το βλέπω εγώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να σχετίζεται με το ποιος μπορεί να κερδίσει από το ταμείο. Ε, είναι περίεργο η πρόταση όλα τα πλοία να πρέπει να πληρώσουν, αλλά μόνο τα ε, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να επωφεληθούν. Ε, πολλά προβλήματα έχει αυτή η πρόταση, αλλά ένα προφανές πρόβλημα είναι ότι ήδη είχαμε κάποιες συγκρούσεις με τους παγκόσμιους εταίρους μας πάνω στις παγκόσμιες μεταφορές. Ό,τι και να κάνουμε λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να είμαστε συνεπείς. Όποιος πληρώνει θα πρέπει να μπορεί να επαφεληθεί κιόλα με κάποιο τρόπο. Επίσης, όπως ανέφερε ο Καρλ, υπάρχει το θέμα της εγκατάλειψης του Ευρωπαϊκού Νεολογίου, διότι αν πούμε μόνο τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε υπάρχει το πρόβλημα της αλλαγής σημαίας και ε, η πρόταση του κυρίου Πρώτη και του κυρίου Ντέιβις ε, μου αρέσουν πιο πολύ διότι ε, καλύπτουν περισσότερο το θέμα αυτό. Τέλος, ε, αλλά εξίσου σημαντικό, θα πρέπει να ε, εξετάσουμε ε, σε ποιες εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο θα επιτρέπουμε τη διάλυση. Εγκαταστάσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός του ΩΣΑ ή οπουδήποτε στον κόσμο αρκεί να είναι φιλική προς το περιβάλλον η εγκατάσταση. Εμένα θα μου άρεσε η τελευταία επιλογή. Παρότι έχω μεγάλο ερωτηματικό στο πρώτο ερώτημα ε, ε, και παρότι νομίζω ότι είμαι καλός πλοηγός, έχω ένα πρόβλημα. Το θέμα είναι η μελέτη αντικτύπου. Δεν είμαστε ίσω οι καλύτεροι να κάνουμε μια μελέτη αντικτύπου, αλλά ποιε θα είναι οι συνέπειε αν επιλέξουμε τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Και ο Κάρλ είπε ότι μόλις λάβαμε αυτή την ε, πρόταση μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, θα την ε, εξετάσουμε. Ναι, αλλά δεν είμαι διατεθειμένος να γράψω ένα κείμενο με βάση αυτή τη νέα έκθεση μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που έχουμε. Δυστυχώς, Έχω την αίσθηση ότι αυτή είναι η μέθοδος που ακολουθούμε όταν ε, δημιουργούμε κακή νομοθεσία. Αυτό που κάνουμε τώρα, λέμε, νομίζουμε ότι έχουμε δύο εξαιρετικέ ιδέες και πρέπει να επιλέξουμε τη μία από τι δύο. Αν χρειαστεί να επιλέξω τώρα, ε, που θα προτιμούσα περισσότερο χρόνο, μάλλον θα έτεινα προ την προοπτική πρώτη Ντέιβις, ένα πρόγραμμα ε, ασφαλιστικού τύπου ή ε, οικονομικών εγγύσεων. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ε, δαπανίσουμε λίγο περισσότερο χρόνο, να εξετάσουμε μήπως υπάρχουν άλλα συστήματα σε άλλους τομείς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ποιε θα είναι οι συνέπειε όσον αφορά τις, τα πλοία που με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ενδιαφερόμενοι τι έχουν πει. Νομίζω ότι πρέπει να πετύσουμε λίγο φρένο. Αν όμω θέλετε να καταλήξετε αυτή τη στιγμή σε ένα συμβασμό, τουλάχιστον να έχετε τώρα κάποιε ενδείξει ποια είναι η θέση μου. Ευχαριστώ πολύ, Κρίστοφ Φιέλνερ. Ο Βιτόριο Πρόντι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το έργο του. Ίσως θα μπορούσε να δουλέψει λιγάκι πιο πολύ τον τομέα της διαφάνειας σε ό,τι αφορά τη διάδοση των απόψεων και των προτάσεων. Ίσως καμιά φορά δεν υπάρχει χρόνος ή δεν υπάρχει διάθεση γι' αυτό. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ήδη ακούστηκαν στη συζήτηση για τον κανονισμό, ιδίω ε, σε ό,τι αφορά τη νομική συμβατότητα του κανονισμού με τις διεθνείς υποχρεώσεις και προηγούμενους κανονισμούς. Όλοι έχουμε διαβάσει ε, τη γνωμοδότηση τη νομική υπηρεσία του, του Κοινοβουλίου. Συγγνώμη. Ίσως κάποιοι δεν διάβασαν την αντίστοιχη γνωμοδότηση του Συμβουλίου που πραγματικά αμφισβητεί αυτή την συμβατότητα. Θα σα υπενθυμίσω ότι η συμβατότητα για την οποία πάντοτε ε, εγώ μιλούσα, αφορά ε, και την ακολουθία ανάμεσα από τον και μεγάλες στρατηγικές ε, ανάπτυξη για την Ευρώπη, όπως η στρατηγική για τις πρώτες ύλε ή η στρατηγική για την αποτελεσματική χρήση των πόρων ή την αρχή του οριπένων πληρώνει ή την αρχή της εκτεταμένης ευθύνης του παραγωγού ή τις αρχές που είναι στη βάση της στρατηγικής μας για τα απόβλητα. Πού ξεχάσαμε αυτή τη, αυτό το σλόγγαν που λέγαμε για την ε, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και εξοικονόμηση. Αν θέλουμε να είμαστε ακόλουθοι σε αυτά που λέμε, θα πρέπει να παραπέμπουμε στη δεσμεύσει που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ενώ Πρόσφατα στην Επιτροπή μας άκουσα την Κομισιόν να καταδικάζει τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία σε απραξία ε, προς όφελος των ασιατικών ναυπηγείων. Μάλιστα, τι είπε αυτό λεξί. Δεν υπάρχει επαρκές δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό πρέπει να αφήσουμε την ανακύκλωση στους Κινέζους ή τους Κορεάτες. Όμως η Βασιλεία μας υποχρεώνει να ανακυκλώνουμε σε οποιοδήποτε ναυπηγείο ή λιμένα που είναι κατάλληλο και βρίσκεται στον ΩΣΑ. Χάθηκαν όλα αυτά τα ναυπηγεία και τα λιμάνια. Εγώ δεν το πιστεύω. Προσπάθησα να βρω μια λύση στο πρόβλημα της αλλαγής ε, σημαίας με ένα εργαλείο που να εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία και να μην αποτελεί, αν θέλετε, ένα νέο φόρο, νέο τέλος ή ένα επιπρόσθετο διοικητικό βάρος. Εν συντομία, εννοώ ένα εργαλείο της αγοράς που να είναι χρήσιμο για όλους και για το περιβάλλον. Ε, και ηρεμήστε, μη φοβάστε, δεν μιλώ για το ETS. Μιλώ για μια ασφάλεια, εξασφάλιση σωστής ανακύκλωσης που να αφορά οποιοδήποτε πλοίο κυκλοφορεί στα ευρωπαϊκά είδωτα και να καλύπτει αν θέλετε τη δαπάνη για την κηδεία τροποντινά του πλοίου σεβόμενη πάντοτε το περιβάλλον σε αναγνωρισμένες και διακριμένες εγκαταστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα συμφωνούσαν ή τουλάχιστον δεν θα είχαν ε, σοβαρό πρόβλημα. Οι ιδιοκτήτες, οι εφοπλιστές ούτε πάλι θα είχαν πρόβλημα. Το πρόβλημα, το πραγματικό, θα ήταν ότι τόσο πολλά πλοία που είναι τόσο παλαιά θα πρέπει άμεσα να ανακυκλωθούν μέσα στην επόμενη πενταετία-δεκαετία. Άρα θα πρέπει να δημιουργήσουμε ad hoc ένα προσωρινό ταμείο που να μας επιτρέψει να ασφαλίσουμε όλα αυτά τα πλοία σε λογική τιμή, όπως προτείνει μία μη κυβερνητική οργάνωση η οποία προτείνει μία παρόμοια λύση με την ασφάλεια. Ε, και ε, είναι αρκετά μακριά από τη λύση ε, που προτείνει ο εισηγητής. Ένας τραπεζικός λογαριασμός ουσιαστικά για την ανακύκλωση. Ίσως θα υπάρξει χρόνος να το συζητήσουμε αυτό το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση των ε, σκιωδών, αλλά πόσο γνωρίζω το Συμβούλιο έχει ήδη αρκετά προβλήματα να επιλύσει πέρα από το θέμα της ασφάλειας δικαίου, ε, που είναι και η ουσία για αυτό τον κανονισμό. Γνωρίζω ότι η Κομισιόν με μια ατχό κομμάδα ομάδα προσπαθεί να χαράξει μια στρατηγική για τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία. Επιτρέψτε μου ότι καλό είναι να δημιουργηθεί ουσιαστικά μια task force για το περιβάλλον, τις επιχειρήσεις, μεταφορές, την απασχόληση, ώστε να δοθεί μια κάποια ελπίδα και στους ανθρώπους και στο περιβάλλον. Σήμερα μάλιστα ε, διαβάζοντας ε, ε, όσο διαμήφθησαν για, σε μια συνάντηση που έγινε για τα ναυπηγεία, βλέπουμε ότι τα στοιχεία είναι καταστροφικά. Έχουν χαθεί άπειρες εργασίες και πιστεύω πραγματικά ότι αν υπάρχουν ναυπηγεία στην Ευρώπη που έχουν την ικανότητα να κατασκευάσουν, να πλοία, ε, μπορούν και να τα αποσυναρμολογήσουν. Αυτό είναι μια εγγύηση ότι θα σεβόμαστε και τους εργαζόμενους και το περιβάλλον. Και αυτό είναι θεμελιώδης εγγύηση που πρέπει να παρέχουμε στους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ, Chris Davis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα χθε ε, ε, τις παρατηρήσεις της κυβέρνησή μου στις τροπολογίες που έχουν καταθέσει οι ευρωβουλευτές σε αυτή την έκθεση. Σπάνια έχω δει τον όρο unwelcome, μη αποδεκτός, ε, τόσους πολλές φορές και αν αυτό αντικατοπτρίζει και την στάση του, Συμβουλίου θα ε-, είναι δύσκολες οι πραγματεύσεις. Όμως ε, όσα αναφέρθηκε, στα όσα είπαν ε, Αυστρία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο και άλλοι για τέτοια ζητήματα. Ο εισηγητής στην έκθεση του αναφέρεται ε, στον ομό καπιταλισμό, αλλά και στην ομή παγκοσμιοποίηση φυσικά, και την ιδέα ότι μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει ένα πλοίο όσο θέλει, μετά μεταφέρει με κάποιον τρόπο τη σημαία. Δεν υπάρχει έτσι καλύτερος τρόπος να το ελέγξει κάποιος αυτό. Και διασφαλίζει ότι πάει προς αποσυναρμολόγηση με την καλύτερη δυνατή τιμή χωρίς ε, κανένα ενδιαφέρον για την υγεία των εργαζομένων ή το περιβάλλον. Οι προτάσει της Επιτροπής γίνονται με καλή πρόθεση βεβαίως και σα ευχαριστώ Επιτροπή. Όμως ε, η βάση είναι η επιτάχυνση της σύμβασης του Χονγκ Κονγκ και πρέπει να γίνουν κάποιες παρατηρήσει για το κατά πόσο πρέπει να υιοθετηθεί ε, η σύμβαση του Χονγκ Κονγκ, αν τον κόπο, γιατί δεν ξέρουμε αν θα επιλύσει όλα τα προβλήματα. Ίσως μπορεί να επανέλθει σε αυτό η Επιτροπή, αλλά ακόμα και αν η σύμβαση ε, του Χοκόν υιοθετηθεί από τον ελάχιστο αριθμό κρατών μελών ή χωρών που πρέπει να το κάνουν, το ζήτημα της ε, σημαίας, του outflagging, δεν ε, καταργείται, δεν σταματά η μεταφορά της σημαίας. Ούτε η προσάραξη ή αποσυναρμολόγηση σκαφών ε, στις ακτές με μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της ε, ρήπανσης. Το πρόβλημα εδώ είναι αυτό ακριβώς, ότι μιλάμε για 90% όλων των σκαφών ε, που όπως νορμολογούνται γίνονται ε, εκτός των κανόνων. Αυτό νομίζω θέλει και ο εισηγητής να αντιμετωπίσει. Εγώ υπέβαλα την τροπολογία 181 για να υπάρχει δηλαδή ένα ταμείο είτε με ρευστό αν θέλετε, είτε με δανεισμό. Ε, βάση για τις υφιστάμενες ευρωπαϊκής νομοθεσίες έκανε αυτή την πρόταση, αλλά μπορώ να την επαναξετάσω. Γιατί υπάρχουν και μειονοκτήματα. Ποιο δηλαδή ελέγχει αυτά τα χρήματα, πώ αντλεί κανεί κεφάλαια από εκεί όταν ε, είναι απαραίτητο πρέπει να εξασφαλιστεί και η στήριξη κοινοβουλευτική για τέτοια ζητήματα και μετά να πούμε σε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν για να μπορεί να σταθεί αυτή η πρόταση και νομικά αλλά και πρακτικά. Και βεβαίως πρέπει να εξετάσουμε και το ζήτημα του κόστους. Ε, όταν λέει ο Κρίστεφερ λοιπόν ότι χρειαζόμαστε αξιολόγηση δικτύπου, έχει δίκιο. Ουσιαστικά λέμε ευχαριστούμε πολύ Επιτροπή. Μας κάνατε μια πρόταση με καλές προθέσεις, αλλά δεν κάνατε τη δουλειά που θέλουμε να γίνει. Το Κοινοβούλιο λοιπόν τώρα προσπαθεί να αδράξει την ευκαιρία να ξαναγράψει την νομοθεσία και να πάρει μια διαφορετική κατεύθυνση, ε, να υποβάλει ε, προτάσεις για να επιληθεί αυτό το ζήτημα μια και για πάντα. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο, να εξετάσουμε το χρονοδιάγραμμα και να μην είμαστε βιαστικοί. Η νομοθεσία αυτή έτσι κι θα έχει πολύ περιορισμένο αντίκτυπο. Δεν νομίζω ότι ε, υπάρχει ανάγκη να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Ας ε, προσπαθήσουμε λοιπόν όσο καιρό για να μας πάρει να καταλήξουμε σε μια πρόταση η οποία να λειτουργεί. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο Πίτερ Φοντάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις ε, για το περιεχόμενο και για τη διαδικασία. Πρόεδρε, επί του περιεχομένου, θεωρώ ότι όλοι θέλουμε να καταργηθεί αυτή η πρακτική της προσάραξης, ε, όπου όλα αυτά τα σκάφη ουσιαστικά ρίχνονται στις ακτές της Ασίας και εμείς θέλουμε να καταργηθεί αυτός ο κίνδυνος του outflagging, με το οποίο χάνουμε μεγάλο τμήμα του στόλου μας. Εδώ όμω θέλουμε και την προαγωγή της ε, απασχόλησης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ε, τόσο υψηλά ποσοστά ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα αυτό επιδεινώνεται και από τις πρακτικές αυτές. Επομένω, έχουμε τρία σημεία επί του περιεχομένου ε, για την κατάργηση ε, του beaching, της προσάραξη, ε, να μειωθεί ο κίνδυνο του ad-flagging και η αύξηση της απασχόλησης. μετά, επί τη διαδικασία. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο από ό,τι έχουμε τώρα. Ήδη βρισκόμαστε στη φάση διαβούλευσης και εξέτασης των τροπολογιών. Εγώ θα ήθελα περισσότερο χρόνο για να εξετάσω αυτά τα τρία ζητήματα με ορισμένου εμπειρογνώμων, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ούτω ώστε να πάρουμε κάποιε απαντήσει πώ μπορούμε να διαμορφώσουμε το καλύτερο δυνατό μοντέλο ε, για να προωθήσουμε αυτά τα τρία ζητήματα. Ιδίω για το τρίτο, το οποίο, το σα ανέφερα, για την απασχόληση. Μήπω, Πρόεδρε, μέσω της ε, συνδρομής από ευρωπαϊκά ταμεία που υπάρχουν ε, να αυξήσουμε την απασχόληση σε αυτό το τομέα. Και μπορώ να θέσω 20 ζητήματα, 20 ερωτήματα γιατί δεν μπορούμε να εξετάσουμε αυτή τη μεταβλητή. Όμως εγώ θέλω να το δω ως μια πρόκληση. Και εφόσον πρόκειται για πρόκληση χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Ανέφερε και ο εισηγητής ε, κάποιες αρχές, αλλά αν θέλουμε ένα πραγματικά καλό πακέτο θα θέλουμε τώρα, πούμε, οι Έλληνες να έχουν ε, ε, τα καλύτερα κίνητρα και τους καλύτερους όρου. Εμείς θέλουμε τον καλύτερο δυνατό πακέτο, του καλύτερους δυνατού όρου. Γι' αυτό ίσως μέσω μιας καλής αξιολόγησης αντικτύπου ή μέσω διατύπωσης των 10 ή 15 βασικών ερωτημάτων και ζητημάτων να... Ε, βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Και δεν θέλω να τσακωθούμε εδώ πέρα, να μαλώσουμε για ε, συγκεκριμένα ταμεία ή από διάφορα επιμέρους ζητήματα. Εδώ ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να βρούμε το καλύτερο δυνατό μοντέλο ε, που επιτυγχάνει και τους τρεις μας στόχους που ανέφερα προηγουμένως. Και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε χρόνο. Να μην περάσουμε ε, κατευθείαν στον πολιτικό διάλογο, χρειαζόμαστε ε, περαιτέρω δουλειά. Ωραία, ευχαριστούμε. Κυρία Βίλτς. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η πρακτική της ε, προσάραξης όσο γίνεται πιο γρήγορα ε, και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να στείλει ένα σεφέ σε μήνυμα ώστε να καταργηθεί η πρακτική αυτή. Δεν μπορούμε να δεχτούμε άνθρωποι στο Μπαγκλαντές ε, να διακινδυνεύουν τη ζωή τους και την υγεία τους για να κερδίσουν οι εφοπλιστές. Ξέρουμε ότι η ναυτιλία είναι διεθνής δραστηριότητα και ότι θα πρέπει να έχουμε γι' αυτό διεθνές καθεστώς. Ε, γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δημιουργήσει οικονομικά κίνητρα ώστε η πρακτική αυτή να γίνει ε, μη ελκυστική για τους ε, ε Ευρωπαίους ε, ε, εφοπλιστές. Η διάλυση των πλοίων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ναυπηγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΩΣΑ. Ε, υπάρχει πρόταση για ε, οικονομικά κίνητρα. Είμαι υπέρ ε, της χρήσης της έρευνας του ΩΣΑ. Το εξή είναι αποφασιστική σημασία. Όλα τα πλοία, όχι μόνο τα πλοία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να συμμετέχουν στο καθεστώ αυτό, ώστε να, υπάρχει, ώστε να υπάρχουν συνθήκε ίσου ανταγωνισμού. Δεν επιτρέπεται να εξωτερικεύουμε τα τοξικά απόβλητα. Ε, και ε, η προσάραξη των ε, πλοίων θα πρέπει να καταλήξει να είναι ένα καθόλου ελκυστικό μέτρο για τους εφοπλιστές. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τον τομέα της ναυτιλίας ώστε να αποφεύγουν στον βαθμό που είναι δυνατόν τις τοξικές ουσίες κατά την κατασκευή των πλοίων. Θέλουμε αποτελεσματική εφαρμογή και έλεγχο και για μένα είναι σαφές ε, ότι θα πρέπει να συμμετέχουν ε, και οι τράπεζες ε, και άλλοι στην λύση. Θα πρέπει να συμμετέχουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αλλιώς ανοίγουμε την πόρτα για οποιαδήποτε απάτη που δεν είναι καθόλου ασυνήθιστη. θα πρέπει μια ε, οποιαδήποτε λύση να έχει ε, ως στόχο να καταστήσει μη ελκυστική την προσάραξη των πλοίων και να ε, αποκατασταθούν οι συνθήκες στις σχετικές χώρες, στις, στις πληγήσεις χώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ οι επόμενοι ομιλητές να περιοριστούν στα δύο λεπτά. παρακαλώ. Εγώ θα σας καλούσα να δείξουμε σύνεση επί του θέματος. Είναι μια παγκόσμια επιχείρηση αυτό το θέμα Προσπαθούμε να επιλύσουμε ουσιαστικά ένα πρόβλημα που συμβαίνει μακριά και έξω από την Ευρώπη. να φέρουμε στην προσάραξη κατά εργασιακά ζητήματα. Και με έναν τρόπο που μάλλον θα είναι αποτελεσματικό. Μια πιο συνετή στρατηγική θα ήταν να προσπαθήσουμε να ε, υιοθετήσουμε το των δυνατών τη σύμβαση του Χονγκ Κόνγκ καθώς αυτό έχει αποδειχθεί το καλύτερο και για την αυτιλία, τον υποκλειστικό κλάδο στο παρελθόν. Όταν μιλάμε για ανθρώπους στο Πακιστάν και τις συνθήκες εργασίας εκεί, τι να σας πω, ξέρετε, στη χώρα μου βλέπω Πακιστανούς που έρχονται να βρουν παρανόμως εργασία στη χώρα μου και κάποιοι μάλιστα κατά τη διέλευση των συνόρων χάνουν τη ζωή τους. Γιατί, γιατί όλα αυτά, γιατί δεν βρίσκουν δουλειά στη χώρα τους και χάνουν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια να μπουν στην επικράτεια. Υπνίγονται στα καράβια που τους μεταφέρουν. Δεν είναι εύκολο να παίρνουν τις αποφάσεις και τη ζωή τους. Δεν ξέρω πόσους τέτοιους έχετε συναντήσει τους τελευταίους μήνες που ήρθαν σε επαφή μαζί σας για το πώς θα νομοθετήσουμε τη ζωή τους τελικά στον Παγκλαντές και το Πακιστάν. Ευχαριστώ κύριε Κροστέτ. Θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ καλή δυνατότητα με αυτόν τον κανονισμό. Συμφωνώ απολύτω με τα όσα υπόθηκαν μόλι τώρα. Έχουμε λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία να αναζωογονήσουμε, αν θέλετε, κάποιους λιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ζητώντας τους να εξειδικευθούν στην ανακύκλωση σκαφών και νομίζω ότι έτσι ρυθμίζουμε και οικονομικά και περιβαλλοντικά και εργασιακά ζητήματα για τους ε, Ευρωπαίους εργαζομένους. Βεβαίως, υπάρχει και η αρχή του ορυπαίνων πληρώνει, δηλαδή οι που είναι, είναι υπεύθυνοι και πρέπει να πληρώνουν. Πρέπει βεβαίω να του τους καλούμε, να του δίνουμε κίνητρα Γι' αυτό να κάνει και αυτό το κείμενο, να ανακυκλώνουν τα σκάφη του στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Για να γίνει αυτό, προφανώς χρειάζεται ένας χρηματοδοτικός ε, οργανισμός, μηχανισμός. Πρέπει να επεξεργαστούμε την ιδέα αυτή ενός ταμείου, στο οποίο θα πρέπει να συμβάλλουν οι εφοπλιστέ. Και αν θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβόλαιο, πρέπει εμείς να καταθέσουμε Προτάσει που να είναι αρκετά επεξεργασμένε, τεκμηριωμένε, ρεαλιστικέ, για να πείσουμε το Συμβούλιο και να προχωρήσουμε. Και στρέφουμε εδώ προ τον εισηγητή. Νομίζω ότι πραγματικά έχουμε μια δυνατότητα, αν θέλουμε, να προχωρήσουν τα πράγματα. Προφανώ 90% ε, τη ανακύκλωση ε, που γίνεται στι χώρε τη Ασία θα πρέπει να σταματήσει, γιατί γίνεται με κακού όρου και πρόκειται για δουλειές που πάνε αλλού. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ξεκινώντας από αυτόν τον κανονισμό, ε, για να αναπτύξουμε την ανακύκλωση στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τις καλύτερες δυνατές ιδέες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο σύντομα στην Κομισιόν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την ε, αρμόδια μονάδα για διαχείριση αμβλήτων στην ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ περιβάλλοντος. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε για τη δουλειά που κάνει η Επιτροπή σας για το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και όπως λέει και η διευθύντριά μου, η Σολέδα Μπλάνκο, που ήταν μαζί σας πριν από κάποιες εβδομάδες, χιλιάδες πλοία αυτή τη στιγμή παροπλίζονται κάθε χρόνο σε απαράδεκτες συνθήκες. Περιβαλλοντικός πώς και κοινωνικός πώς. Καθώς ε, ε, προσαράσουν στις ακτές της ε, Νοτιοανατολικής Ασίας. Μιλήσατε ειδικά για τα οικονομικά κίνητρα και τους μηχανισμούς ασφάλισης. Σε ό,τι αφορά την, ε, τις ασφάλειες, ε, θα έλεγα ότι είναι κάπως ε, αμήχανη θέση μας και μεικτά τα συναισθήματα, διότι τρέφουμε κάποιες σοβαρές αμφιβολίες στην Κομισιόν θα έλεγα. Σε ό,τι αφορά τον διοικητικό αντίκτυπο και το πώς θα διαχειριστούμε το βάρος οποιοδήποτε τέτοιου οικονομικού κινήτρου. Ανάμεσα στις επιλογές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, η ασφάλεια φαίνεται να είναι ένα από τα λιγότερα επαχθή εργαλεία. Όμως συμφωνούμε και εμείς μαζί σας. Ο μηχανισμός αυτός δεν είναι κατάλληλα σχεδιασμένος για να επιτύχει τον στόχο που εσείς επιθυμείτε. ο οικονομικός μηχανισμός τύπου ασφάλεια έχει σκοπό να προστατεύσει τους πλειοκτήτες από κινδύνους που δεν μπορούν να ελέγξουν. Σε αυτή την περίπτωση, ο κίνδυνος δημιουργείται από την ίδια την απόφαση του πλειοκτήτη. Θεωρούμε λοιπόν ότι η επιλογή της ασφάλειας δεν είναι ο κατάλληλος μηχανισμός για αυτό το ζήτημα. Και θεωρούμε ότι δεν είναι επιχείρημα ότι η λύση της ασφάλειας είναι μια πιο απλή λύση από άλλες, διότι δεν μας καλύπτει ε, εν προκειμένου. Ε, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να πω κι εγώ ότι και εμεί στην Κομισιόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα θεμελιώδες δίλημα. Κάποιοι ε, από εσά το έθιξαν ήδη. Είναι μια επιλογή ανάμεσα στην εφαρμογή οικονομικού κινήτρου για ευρωπαϊκά πλοία μόνο ή και για τα άλλα πλοία. Ένα δίλημα με δύσκολη λύση. Ό,τι τελικά και εσείς επιλέξετε να κάνετε, τελικά θα βρείτε μπροστά σας περίπλοκα πολιτικά προβλήματα, ειδικά αν επιλέξει την επιλογή που θα καλύπτει μόνο τα ευρωπαϊκά πλοία. Και ουσιαστικά θα παρέχετε κίνητρα για την επιλογή άλλων ε, μειογνωμόνων έξω από την Ένωση. Κάτι άλλο που θέλω να επισημάνω είναι ότι η Κομισιόν ενέταξε στην ανάλυση που έκανε και την εναλλακτική εκείνη που προβλέπει ένα οικονομικό μηχανισμό πριν σας υποβάλουμε την νομοθετική μας πρόταση. Το σκεφτήκαμε, το αναλύσαμε αυτό. Κάναμε και τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Και καταλήξαμε τελικά ότι η καλύτερη επιλογή θα ήταν ένα ισχυρό αποτρεπτικό σύστημα, ένα σύστημα κυρώσεων προς τους πλοκτήτες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ε, συμμόρφωσης εννοώ με το καθεστώς ανακύκλωσης. Μιλώ για κυρώσεις προς τους πλοκτήτες. Αυτό θα είναι αποτρεπτικό, θεωρούμε. Ένα ισχυρό αποτρεπτικό κίνητρο, ε, πιο ισχυρό από ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Δώσω το λόγο στον εισηγητή να απαντήσει. Ευχαριστώ. Ο κ. παράλληλα και ο κ. Κρυστέιβη συνόψισαν το θέμα. Δεν ναι, θέλουμε αυτούς τους στόχους. Θέλουμε μια καλή μεταχείριση για αυτά τα σκάφη. Θέλουμε ένα σύστημα που να είναι αποτελεσματικό. Εμείς ε, όμως πρέπει να να πιστέψουμε ειλικρινά στην λύση που θα επιλέξουμε. Να είναι μια περίπτωση που όλοι μας έχουμε παρόμοιους στόχους. Δεν ξέρουμε όμως πώς να τους επιτύχουμε. Και όταν λέω πρέπει να είμαστε γρήγοροι, δεν εννοώ να βιαστούμε και να φάνουμε ανόητοι. Πρέπει να τα κάνουμε σωστά τα πράγματα. Κρίστοφερ. Υπάρχει μελέτη δικτύπου και σε 6 Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί και επισήμως. Η μελέτη δικτύπου θα μας βοηθήσει πραγματικά να επιλέξουμε να στις λύσεις. Ε, δεν είναι ένα θέμα ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Θα πρέπει να μελετήσουμε πρακτικά ε, όλα τα υπέρ και κατά και χρειαζόμαστε μια κάποια καθοδήγηση. Έπειτα, πρέπει να βρούμε μια λύση, αλλά μια λύση αποτελεσματική. Κύριε Σκυλακάκη, η σύμβαση Hong Kong, ακόμα και αν την εφαρμόσουμε, ξέρουμε ότι θα είναι κάτι χρονοβόρο στη δικασία, αλλά και να το κάνουμε, δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Δεν είναι αρκετά ισχυρή. Βλέπετε ότι η Κομισιόν προσπαθεί στην πρότασή τη να καλύψει τα κενά και τα προβλήματα που έχει η σύμβαση του Χοκόγκ. Αυτό που κάνω και εγώ. Ας προσπαθήσουμε να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα στην Ευρώπη και αν τελικά τα καταφέρουμε αυτό να επηρεάσει και εκτός Ευρώπης, καλό είναι και αυτό. Γιατί τα κάνουμε όσα κάνουμε τώρα. Διότι είναι συνέπεια της κατανάλωσής μας όλο αυτό το πρόβλημα. Έχουμε συνέπειες που σκοτώνουν ανθρώπους, σκοτώνουν το ίδιο το περιβάλλον σε διάφορα μέρη του κόσμου. Κρίς. Ναι, η Βρετανική κυβέρνηση ε, δεν βλέπει καθόλου θετικά την πρότασή μα. Αλλά δεν έχω έρθει σε επαφή με την Βρετανική κυβέρνηση. Όμω έχω έρθει με άλλου. Κανένα δεν είπε ότι δεν πιστεύω σε ένα χρηματοδοτικό μέσο. Όλοι λένε, Α, ενδιαφέρουσα πρόταση για να δούμε πώ θα μπορούσε να λειτουργήσει. Κανένα δεν είπε όχι κατηγορηματικά. Αν λοιπόν επιτύχουμε να ολοκληρώσουμε ε, επιτυχώς αυτό το φάκελο. Αν χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας, μπορούμε κάτι να καταφέρουμε, πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά δεν είναι και αδύνατο, δεν θα είναι και θαύμα. Ε, Εντάξει, σα καταφέρουμε να φανούμε και λίγο εφάνταστοι εδώ στο Κοινοβούλιο. Ζητώ συγγνώμη ε, κύριε Υπουργέ που έχω καταχράσει το χρόνο σα. δεν θα ξαναπώ μετά τη δεύτερη φορά τέτοια λόγια, οπότε έχω καλυφθεί. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Καρλ Σλίτερ, 19 Φεβρουαρίου μάλλον θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας, ε, αλλά θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε διότι δεν είναι ακόμα βέβαιο. Έχουμε ικανό ε, εισηγητή είναι και λίγο ε, σκεπτικός. Ε, δεν, δεν έχουμε ακόμα ημερομηνία ε, και για την Ολομέλεια ακόμα. Έτσι περνάμε στον επόμενο μιλητή. Καλωσορίζουμε τον Ιρλανδό Υπουργό Περιβάλλοντος. Κοινοτικής και τοπικής αυτοδιοίκησης της Ιρλανδίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο συνδυασμός αυτός. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Φιλ Χόγκαν. Είχαμε και στο παρελθόν επαφές με την Προεδρία και το ζήτημα που μόλις συζητήσαμε ελπίζουμε ότι και αυτό ε, θα προωθηθεί από εσά στο Συμβούλιο. Έχουμε και κάποια άλλα σημαντικά θέματα. Καταρχήν, Έχουμε τις δημοσιονομικές προοπτικές, ε, όπου, όπου εμπίπτει το πρόγραμμα LIFE, εμπίπτουν τα προγράμματα LIFE, αλλά και η μελλοντική γεωργική πολιτική. Είχαμε σήμερα ε, σχετική ψηφοφορία, συζητήσαμε με τους συναδέλφους μας από την ε, Επιτροπή Γεωργίας και η δική μας γνωμοδότηση προβλέπει διαφορετική κατεύθυνση. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε τι μορφή πώς μάλλον θα αντικατοπτρίζεται η μεταρρύθμιση της γεωργίας στην πολιτική. Επίσης έχουμε ε, τις οριακές τιμές για τα αυτοκίνητα μέχρι το 2020 και Έχουμε επίσης και μία έκθεση την οποία έχω την ε, τιμή να εκπονώ ε, που έχει να κάνει με την προστασία του, περιβάλλ... του κλίματος και το λεγόμενο backloading. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών νομίζω ότι λειτουργεί καλά, αλλά θα μπορούσε να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα. Διότι πρέπει να έχει συγκεκριμένη τιμή το διοξείδιο του άνθρακα. Αύριο θα έχουμε τη σχετική συζήτηση εδώ. Αλλά θα ήθελα πολύ να ακούσω πώς προσεγγίζει το θέμα αυτό το Συμβούλιο. Ώστε τελικά τον Μάρτιο να μπορέσουμε να κλείσουμε το θέμα αυτό. Τον Φεβρουάριο θα έχουμε σχετική ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή μας ε, και τον Μάρτιο θα λάβουμε την ε, τελική απόφαση. Πολλά θέματα λοιπόν θα εξατεστούν μέσα στο επόμενο εξάμεινο, πολλά θέματα πρέπει να κλείσουμε μέσα στο επόμενο εξάμεινο και τα προγράμματα δράσης για το περιβάλλον, αλλά ε, και μελέτες αντικτύπου ε, στο, για το περιβάλλον, καθώς ε, και το e-look, η έμεση χρήση εκτάσεων. Κύριε Χόγκαν, λοιπόν, και το Συμβούλιο έχει πολλή δουλειά να κάνει, δεν θα βαρεθούμε νομίζω καθόλου. Σας δίνω τώρα τη δυνατότητα μέσα σε 10 λεπτά να μας παρουσιάσετε τα ε, βασικά θέματα για σας. Και κατόπιν θα έχουν τη δυνατότητα οι συνάδελφοι να θέσουν ερωτήσεις. Πρώτα θα δώσουμε το λόγο στους συντονιστές και κατόπιν στους άλλους συναδέρφους. Έχετε το λόγο. Περιμένουμε να ακούσουμε με χαρά αυτά που έχετε να μας πείτε. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα μαζί σα για να σα περιγράψω αυτό που εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ φιλόδοξη περιβαλλοντική ατζέντα για την 7η Ιρλανδική Προέδρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ στο Κοινοβούλιο. Μετά τον ε, διορισμό μου πριν από δύο χρόνια, ε, είχα δηλώσει ότι η συνεργασία με το Κοινοβούλιο είναι σημείο προτεραιότητας για τι προετοιμασίε της Προεδρίας, αναγνωρίζοντα τον κεντρικό ρόλο του Κοινοβουλίου στη δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, από τον Οκτώβριο του 2011, όπου ξεκίνησα τη συνεργασία με τα μέλη της επιτροπή ε, συνεχίζουμε από τότε με πολλέ ε, συναντήσει, όπω και σήμερα, στι Βρυξέλλες αλλά και στην ε, συνδιάσκεψη για το κλίμα στην Τόχα τον προηγούμενο μήνα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εσένα Ματίας και όλα τα μέλη της Επιτροπής που έχω συναντήσει που ε, δώσατε λίγο από τον χρόνο σας, εμένα και στην ομάδα μου. Γιατί το υψηλό επίπεδο δέσμευση ε, για τη συνεργασία μα είναι απαραίτητο στοιχείο για την ε, επιτυχή εξέλιξη των διαπραγματεύσεων στου επόμενου μήνε. Όπω ξέρετε, η Ιρλανδική Προεδρία λαμβάνει χώρα σε μια ε, οικονομική συγκυρία γεμάτη προκλήσεις. Ε, μια περίοδο που δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε ε, στα συνηθισμένα, στο μοντέλο που υπήρχε πριν από την κρίση. Ωστόσο, μέσω της στρατηγικής Ευρώπη 2020 έχουμε σημαντικούς δείκτε. ε, στρατηγικής εξέλιξης όπως η οικοδόμηση μιας έξυπνης, ευφυούς Ευρώπης, βιώσιμης Ευρώπης και Ευρώπης χωρίς αποκλεισμού. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να εστιαστούμε στην ε, σταθερότητα, στις ε, θέσεις εργασίας και στην ανάπτυξη, στην καινοτομία, αλλά και στην ενσωμάτωση των αρχών της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας σε όλες τις πολιτικές, σε όλους τους πολιτικούς τομείς, και το εξαμήνου. Αυτά τα θέματα διέπουν το σύνολο του, ευρωπαϊκού, του Ιρλανδικού προγράμματος βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού μας θεματολογίου, ε, κυρίως ό,τι αφορά την διαμόρφωση μιας ε, Ευρώπης με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα και αποδοτικότητα σπόρων. Σήμερα θέλω να σας παρουσιάσω συνοπτικά το ε, πρόγραμμα της Ιρλανδικής Προεδρίας από την περιβαλλοντική σκοπιά, αλλά και τα βασικά στοιχεία της διεθνούς μας ατζέντας σε ό,τι αφορά τη στρατηγική, το 7ο πρόγραμμα δράση για το περιβάλλον είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία για την ε, Προεδρία μα, Είναι ένα από τα κύρια σημεία ε, στον περιβαλλοντικό τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και θα θέσει σε ισχύ βασικά στοιχεία της στρατηγικής Ευρώπης 2020. Πολλά έχουν γίνει τους τελευταίους ε, μήνες ε, για αυτή την πρόταση και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Κυπριακή Προεδρία ε, για το έργο της αυτό το φάκελο. Καθώς είχαμε έξι συνεδριάσεις ομάδας εργασίας κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο μηνών, έχουμε έναν φιλόδοξο στόχο να φτάσουμε στην πρώτη ανάγνωση πριν από το τέλος της Προεδρίας. Και προσβλέπω σε συνέχιση της συνεργασίας μας με το Κοινοβούλιο. Το άλλο βασικό στοιχείο της περιβαλλοντικής στρατηγικής στο οποίο θα επικεντρωθούμε είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική προσαρμογή ε, στο κλίμα. Εάν δημοσιοποιηθεί αυτή, δημοσιευθεί μάλλον η πρόταση από την Επιτροπή το Μάρτιο ή Απριλίο, ε, εμείς θα, θα το ορίσουμε ως βασική προτεραιότητα. Μετά, Υπάρχουν πολλέ νομοθετικέ προτάσεις μπροστά μας. Ε, δεδομένων των περιορισμών σήμερα θα εστιαστώ στι βασικές για μα ε, προτάσεις. Ε, κυρίως ό,τι αφορά το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν δύο σημαντικές προτάσεις για, την, ε, για τις εκπομπές εξουδίου του άνθρακα από τα νέα αυτοκίνητα και φορτηγά. Μετά έχουμε δύο τροπολογίες του ε, προγράμματος του εμπορίας εκπομπών ε, το πρώτο, η πρώτη από τις τροπολογίες αυτές, τις τροποποιήσεις μάλλον, αφορά ε, ε, την ε, επιπρόσθετη νομική ασφάλεια και η δεύτερη αφορά την ναυσιπλοεία, συγγνώμη, την αεροπλοεία. και αυτή συνδέεται με το πρόγραμμα εμπορίας εκπομπών. Και πάλι σκοπεύουμε να επιτύχουμε πρώτη ανάγνωση και σε αυτή την πρόταση. Υπάρχει μια σειρά νομοθετικών προτάσεων στον τομέα του κλίματος που δεν θα ε, καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε, ωστόσο θα... Ε, είναι και αυτές οι προτεραιότητες για μας. Δύο είναι οι βασικές προτάσεις. Πρώτον, να αυξηθούν οι, προσπάθειες να μειωθούν κάποιες ε, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και φθοριούχων μάλιστα, ε, Εξαιτία των περιβαλλοντικών τους ε, επιπτώσεων. Δεύτερον, ε, η έμεση αλλαγή της χρήσης γης. Παρότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα πολιτικά και τεχνικό, θέλουμε να έχουμε μια συζήτηση προσανατολισμού στο Συμβούλιο του Μαρτίου και μετά να έχουμε και μια έκθεση πρώτου τον Ιούνιο που θα παραδώσουμε στη Λιθουανική Προεδρία. Και πάλι σε ό,τι αφορά τους νομοθετικούς φακέλους σε επίπεδο περιβάλλοντος και πάλι έχουμε υψηλό επίπεδο ε, φιλοδοξία σε ό,τι αφορά τις βασικές ουσίες ε, στο νερό. Θα εργαστούμε μαζί σας για να υπάρξει συμφωνία πρώτης ανάγνωσης. Δεύτερη πρόταση, αυτή που μόλις συζητήσατε για την ανακύκλωση σκαφών, ε, ούτω ώστε όλα τα σκάφη να ανακυκλώνονται με έναν τρόπο που θα προστατεύει την υγεία των εργαζομένων αλλά και το περιβάλλον ε, από τους ε, κινδύνους κάποιων πολύ κακών πρακτικών σε αυτόν τον τομέα. Και εδώ ελπίζουμε να επιτύχουμε πρώτη ανάγνωση. Σε ό,τι αφορά τις οδηγίες για τις ε, μπαταρίες, ε, για να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή με την χρήση ορισμένων επιπέδων καδμίου, έχουμε ως στόχο και πάλι να υπάρξει πρώτη ανάγνωση. Τώρα, για την πρόταση LIFE, πρέπει να χαιρετήσουμε την σημαντική πρόοδο που επέτυχε η Κυπριακή Προεδρία. Συνδέεται με το στο νομικό πλαίσιο βεβαίω μέχρι το 2020. Γι' αυτό και θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ τι εξελίξει σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχει πρόταση από την Επιτροπή για κανονισμό για την ε, πρόσβαση και επιμερισμό των ωφελών για τους γενετικούς πόρους. Ε, για την κύρωση του πρωτοκόλου Ναγκόια που δίνει πρόσβαση ή ρυθμίζει την πρόσβαση στις, στους παραδοσιακούς γενετικούς σπορούς, ιδιαίτερα στον απτυσσόμενο κόσμο και πώς τα ωφέλη αυτά από αυτούς τους σπορούς θα πρέπει να καταμερίζονται ε, ανάμεσα στις ε, ε, χώρες που τις παρέχουν και στις τοπικές κοινότητες. Μάλλον δεν θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες αυτού του Βακέλου κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, όμως θα έχουμε μία συζήτηση προσανατολισμού το Συμβούλιο, στο Συμβούλιο το Μάρτιο και μετά έκθεση προόδου, προόδου τον Ιούνιο. Τέλος, τελευταία νομοθετική πρόταση είναι η μεταρρύθμιση της οδηγίας ε, για την ε, ε, έκθεση περιβαλλοντικού αντικτύπου. Είναι σημαντική και περίπλοκη πρόταση και θα μας πάρει χρόνο να την προωθήσουμε και πάλι το ίδιο με τα προηγούμενα, συζήτηση προσδολισμού το Μάρτιο και έκθεση προόδου τον Ιούνιο. Παρότι τα ζητήματα, τα πυρηνικά και της ε, ακτινοβολίας είναι κάτι το οποίο εξετάζει το Συμβούλιο Ενέργειας, ε, η, εθνική πολιτική ευθύνη παραμένει στο δικό μας ε, Υπουργείο. Ε, θα εξετάσουμε λοιπόν ως προς αυτό την ε, οδηγία βασικών προτύπων ασφαλείας που αποτελεί προτεραιότητα για μας γιατί διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των εργαζομένων, μέλων των πολιτών και ασθενών και αφορά νέες ε, ε, διατάξεις για την ε, καταγραφή κάποιων ραδιενεργών υλικών. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά την διεθνή περιβαλλοντική ατζέντα και θεματολόγια, εδώ έχουμε πέντε τομείς προτεραιότητας. Πρώτον, ε, τι συμβαίνει με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, ε, των οποίων ηγείται το, το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ε, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένους ουσίες. Έχουμε διαπραγματεύσει το τελευταίο ε, το τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων στη Γενέβη την τελευταία εβδομάδα και η Ιρλανδική Προεδρία πρέπει να πω ότι έπαιξε σημαντικό και θετικό ρόλο στη διαδικασία και υπήρξε και συμφωνία το προηγούμενο Σάββατο. Η συνέχιση του Ρίο θα είναι άλλη προτεραιότητα για μας ε, συνεχίζοντας από τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, θα έχουμε και πάλι, θα διδραματίσουμε ηγετικό ρόλο στη διαχείριση της ε, Συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 23η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της UNEP που θα λάβει χώρα τον επόμενο Σεπτέμβριο. Και από πλευρά ανάπτυξη βεβαίω θα συνεργαστούμε με τους συναδέλφους ε, για να προαγάγουμε τους ε, αναπτυξιακούς στόχους της χιλιατηρίδας. Ε, τον Μάρτιο συνεχίζουμε στο διεθνές κοινικό με το site Scope στη Bangkok για, συγκεκριμένα, για τη διατήρηση συγκεκριμένων ζωικών ειδών όπως ο αφρικανικός ελέφαντας, ρινόκερος και το καθεξής. Οι ευρωπαϊκέ προτάσει που θα συζητηθούν είναι βασική προτεραιότητα για μα, ό,τι αφορά ένα ε, συγκεκριμένο είδο ε, ε, καρχαρία υπό εξαφάνιση. Άλλη σημαντική προτεραιότητα θα είναι οι προβολτικέ πτυχέ των τριών συμβάσεων του ΟΗΕ για τα απόβλητα και τα χημικά στο Χόλμη, Ρότερνταμ και Βασιλεία. Τον Απρίλιο και τον Μάιο θα λάβει η χώρα συνδιάσκεψη στην Γενέβη για αυτό το θέμα και εκεί θα δούμε πώς η διεθνή διακυβέρνηση μπορεί να βελτιωθεί για καλύτερη συνεργασία και συντονισμό. Τέλος, Πρόεδρε, από διεθνούς πλευράς υπάρχει βεβαίω ένα κρίσιμη σημασία ζήτημα για τις ε, διεθνείς κλιματικές διαπραγματεύσεις υπό το, ε, τη Σύμβαση Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ. Ενώ υπήρχε πρόοδο και στην ΕΝΤΟΧΑ τον προηγούμενο μήνα, αλλά και το για το 2015 θα συνεχιστεί όλη αυτή η ε, διαδικασία ε, με τα 195 μέρη που υπογράφουν τη σύμβαση για την μείωση των εκπομπών ε, αερίων του θημοκηπίου. Εφόσον οι υπογράφοντες έχουν μια νέα δέσμευση και καλύπτουν μόλις το, όμως το 15% των εκπομπών, είναι πολύ σημαντική αυτή η συνολική συμφωνή του 2015 και η Ιρλανδική Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί, ιδιαίτερα στι συναντήσει τη Βόνη ε, τον Απρίλιο, Μάιο και τον Ιούνιο. Ε, να σα ενημερώσω και για το άτυπο Συμβούλιο 22-23 Απριλίου στο Δουβλίνο για να δούμε πω η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διδραματίσει το δικό τη ρόλο στι διεθνεί κλιματικέ διαπραγματεύσει. Ε, Βεβαίω, ανάλογα και με την ολοκλήρωση του έργου από την Επιτροπή, θα εξετάσουμε τα επόμενα βήματα για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το άτυπο συμβούλιο θα αποτελέσει και μια ευκαιρία για χρήσιμες συζητήσεις ε, για την ενιαία αγορά για τα βιολογικά προϊόντα ε, και για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και το αστικό περιβάλλον. Θα έχουμε και μια κοινή συζήτηση με τους ε, Υπουργούς Ενέργειας και σας έχω ήδη προσκαλέσει, Πρόεδρε, να συμμετάσχετε σε αυτή την συνεδρίαση. Σας προσκαλώ και στην και στο κάστρο του Δουβλίνου για αυτή την ε, συνάντηση που έχει λάβει και διπλή πιστοποίηση μάλιστα για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τέλος, έχουμε, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε πολλές προτεραιότητες ε, στο στρατηγικό μας θεματολόγιο ε, που μας δίνει τη δυνατότητα να αφήσουμε και τη δική μας ασφραγίδα στα γεγονότα, που είναι και ένα από τα βασικά ωφέλη της ε, ε, εκπεριτροπής προεδρίας. Έτσι λοιπόν ακολουθούμε με διάφορες εμβληματικές πρωτοβουλίες όπως είναι η Ευρώπη 2020 και το 7ο EAP ε, με αποδοτικότητα πόρων και με το βλέμμα στραμμένο προς τη δράση. Και βέβαια πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέχρι τον ορίζοντα 2020 που τώρα απέχει λιγότερο από 8 χρόνια. Οι νομοθετικέ μας προτάσεις είναι κρίσιμη σημασία σε ό,τι αφορά τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα σε πολλούς τομείς ε, και η δυνατότητα πρώτη ανάγνωση ε, θα δοθεί μόνο αν υπάρχει καλή και αποδοτική συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ενεργό ρόλο ε, και υψηλό επίπεδο δέσμευσης με ε, όλο τον ε, κόσμο. Επομένω ε, ε, το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, με αισιοδοξία, αλλά και με διάθεση για δουλειά, για βιώσιμη ανάπτυξη, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και βιωτικού επίπεδου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τι ε, μεμονωμένες ε, προσπάθειε Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και επιτροπή, αλλά και από τη συνεργασία μεταξύ αυτών των ε, θεσμικών οργάνων. Για μένα είναι μια προτεραιότητα εδώ και 15 μήνε να προετοιμάσω το έδαφο για την Προεδρία μα μέσω επικοδομητικού διαλόγου με σένα, Προεδρέ, και με τα μέλη τη Επιτροπή και με του εισηγητέ και με του σκιώδει. Και θα βρίσκομαι σε επαφή μαζί σα Καθώ οι τα θα εντατικοποιούνται μέσα στου επόμενου μήνες. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Έχουμε πολλή νομοθεσία υπό Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στους συντονιστές και θα μιλήσω γερμανικά. Έχουμε και ακροατές εδώ σήμερα άνθρωπους, επαγγελματίες που εφαρμόζουν καθημερινά την ε, ε, νομοθεσία μας ε, από την περιοχή Ρουρ. Έχουμε τον Δήμαρχο και δημοτικού συμβόλου. Δυστυχώ δεν επιτρέπει να σα δώσω το λόγο, αλλά καλώ ήρθατε και χαιρόμαστε που συμμετέχετε στη συνεδρίασή μα. Περνάμε λοιπόν στον πρώτο γύρο. Διαβάζω τα ονόματα των συντονιστών που θα πάρουν το λόγο για να βεβαιωθώ ότι δεν ξέχασα κάποιον. Dann kommt Joe Lein, dann Chris Davis, Bas Eichhaut, Christa Klaas, Karl-Heinz Florenz, François Grosset, dann der Kollege Gebrandi und abschließend Karl Schlüter und Corinne Lepage. Και τέλος ο Καλ Σλίτερ, η Κορίν Λεπάζε και η Μαρκαρέτα Ουλσκog. Και ο Βικτόριο Πρόντι. Κλείνω τον κατάλογο των ομιλητών. Δύο λεπτά ο καθένας, διότι θα ήθελα να δώσω σε όλους το λόγο. Ο Ρίχαρτ Σέιμπερ πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Χόγκαν έχει ε, ένα ε, πολύ ευρύ πρόγραμμα πρωτοβουλειών. Αναφερθήκατε στο σύστημα εμπορία εκπομπών και ε, το backloading. Μήπω μπορείτε να μας, πείτε σύντομα πώς έχει η κατάσταση στο Συμβούλιο. Ε, πρόκειται να ψηφίσουμε πάνω στην έκθεση αυτή. Και υπάρχουν κάποιες προτάσεις που πρόκειται να απορριφθούν λόγω νομικής βεβαιότητας και και επειδή ε, δεν είναι σκόπιμες για την επίτευξη του, του στόχου της μείωσης που θέλουμε. Ε, υπάρχουν ε, θέματα στα οποία δεν έχουμε δώσει την απαραίτητη προσοχή. Έχουμε Υπάρχουν ε, διάφορα αέρια και τα λοιπά τα οποία θέλουμε να ε, απαγορεύσουμε μακροπρόθεσμα ε, και να εφαρμόσουμε την απαγορεύση αυτή. Υπάρχει το θέμα του ύδατος και των διαφόρων ουσιών. Μήπως μπορείτε να μας πείτε πώς η Ιρλανδική Προεδρία θέλει να διασφαλίσει να μπορέσουμε με τα φάρμακα να περάσουμε σε πράσινη κατεύθυνση. κατεύθυνση. Νομίζω θα είναι ενδιαφέρον για το δήμαρχο του, της περιοχής Ρουρ ε, να ακούσει πώς έχετε σκοπό να αφαιρέσετε τις επικίνδυνες ουσίες ε, από ε, τα υγρά απόβλητα και να μας πείτε πώς ακριβώς βλέπετε το όλο θέμα αυτό. Τέλος, ε, όσον αφορά την ποιότητα του αέρα. Αυτό είναι πρόβλημα στη Γερμανία σε πολλές πόλεις. Ήδη έχουμε φτάσει τα οριακά επίπεδα. Προβλέπετε εδώ περαιτέρω... προβλέπετε πιο αυστηρή ε, νομοθεσία, διότι και η Γερμανία και η Αυστρία έχουν σοβαρά προβλήματα στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Ρίχαρ Ζέμπερ. Ο Γιώλα είναι δύο λεπτά. Ε, κύριε Προεδρεύοντα, σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας. Ε, ακούγονται πολύ καλά αυτά που προτείνετε. Ε, ελπίζω η Ιρλανδική Προεδρία να ε, μείνει στην ιστορία ως πράσινη Προεδρία. Έχουμε δει πολλές προεδρίες. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Είχαμε τη, την διάσκεψη του Ρίο, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε διάφορα ε, διάφορες υποχρεώσεις ε, μεταξύ άλλων ε, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τα SDGs. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι απέγινε η δική μας στρατηγική βιωσιμότητα, που υιοθετήθηκε το 2001, έληξε το 2012 και εξαφανίστηκε. Τώρα, στο πλαίσιο της αναβίωσης ε, του Ρίο, θα πρέπει εσείς να ζητήσετε αναβίωση της ε, πολιτικής βιωσιμότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επίσης, όσον αφορά το ε, UAP είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε πολύ να το δούμε να ε, διέπει και άλλες πολιτικές. Ενδιαφέρον θα είναι να ε, ε, συναντηθεί το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος με το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, διότι εμείς θέλαμε τρεις στόχους μέχρι το 2030 και όχι έναν χρειαζόμαστε και για την ε, βιομηχανία, συγκεκριμένο στόχο για την ε, βιομηχανία όσον αφορά ε, το, το περιβάλλον και επίσης Όσον αφορά την προστασία του εδάφους, πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο το χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη, που είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε προπολού να έχουμε λύσει. Και επίσης, ε, όσον αφορά, και επίσης μας ενδιαφέρει και η εφαρμογή της ε, στρατηγικής ε, φτωχή σε διοξίδιο του άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώ. Επόμενο είναι ο Κρι Ντέιβι. Um, Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομο. Δύο σχόλια. Από τη στιγμή που ανάλευε η Ιρλανδία την Προεδρία, οι τιμέ του άνθρακα έπεσαν στο ελάχιστο. Ε, ελάχιστη τιμή ρεκόρ. Εσείς φταίτε γι' αυτό. Ναι, είπατε ότι υπάρχει πρόταση του backloading. Και είναι μια πρόταση που πιστεύω ότι έχει σκοπό να διατηρήσει ένα μηχανισμό της αγοράς που αυτή τη στιγμή ε, κινδυνεύει να καταρρεύσει. Δεν ξέρω ακριβώς ε, τι προτείνετε να κάνετε το Συμβούλιο. Δεύτερον, για το site Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Στις διασκέψεις ΆΙΤΙΣ η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά παρουσιάζεται ως μια ομάδα κρατών μελών. Δηλαδή υπάρχει συντονισμός, αλλά δεν υπάρχει ενιαία Εγώ θέλω να επισημάνω ότι χρειάζεται τέτοιο συντονισμό για να μπορούμε να έχουμε ισχυρή θέση. Δεν υπάρχει χειρότερο από το να ακούς ότι τελικά απέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποια ζητήματα γιατί δεν μπορούν οι εταίρετες να συμφωνήσουν. Thank you very much, Chris. Next speaker is Bas Eichert. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την παρουσίαση του προγράμματο για το επόμενο εξάμενο και εγώ προσβλέπω συνεργασία μαζί σα για κάποια από τα ζητήματα που θα σα απασχολήσουν. Έχω να πω λίγα λόγια για το ETS και για τι ε, ε, ενεργειακέ πολιτικέ περιβάλλοντο. Για το ETS, είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα στο Συμβούλιο. Μια χώρα πρέπει να πείσετε, τη Γερμανία. Υπ' αυτή την έννοια, εστιάζω το ερώτημά μου ω το εξή πώ τελικά θα κερδίσετε τη Γερμανία και πώ θα εξηγήσω στον Πίτερ Μάιερ ότι ένα συμβιβασμό που οδηγεί στην εποχή ουσιαστικά είναι άρνηση. Αναρωτιέμαι ποια θα είναι η στρατηγική σα και ε, στις συναμιλίες με τον Πίτερ Μάιερ και έπειτα για το backloading, όπως είπε και ο Κρις. Πέρα από αυτό χρειαζόμαστε διαφορετικά μέτρα πώς θα προωθήσετε αυτό το διάλογο βελτιώνοντας τα θεωρητικά μέτρα για το ETS. Ε Ιδάλλως θα υπάρχει πρόβλημα και σε δύο χρόνια και με το ETS. Ε να περάσω τώρα στη διεθνή σκηνή για το κλίμα. Κατανοώ ότι στις 22 και 23 Απριλίου έχετε ένα άτυπο συμβούλιο. Όμως για την Ευρώπη ο χρόνος ε, κινδυνεύει να εξαντληθεί. Ο Μπάλκι Μούν είπε στην Τόχα ότι θα καλέσει τους διεθνείς ηγέτες να συνέλθουν το Σεπτέμβριο του 2014 με θέμα πώς θα γεφυρθεί το χάσμα των δύο βαθμών και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και που δεν αρκούν ήδη ε, κάποιοι ε, έχουν δεσμευτεί για μείωση των εκπομπών κατά 30%. Εμείς έχουμε δεσμευτεί για 20%. Πώς μπορείτε να αγγιηθείτε ότι τελικά η Ευρώπη ένα χρόνο μετά το δικό σας τύπο συμβούλου θα μπορούσε να επιτύχει περισσότερα. Ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας ευρωεκλογέ που είναι μια χαμένη χρονιά ουσιαστικά. Όμως ο, ο κόσμος περιμένει να ηγηθείτε. Το ίδιο είχε το 2015. Την επόμενη χρονιά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη για ένα πακέτο με το 2020. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το δικό σου εξάμεινο με μεγάλη, αν θέλετε, μαεστρία, δεν θα μπορέσουμε ε, να είμαστε ούτε έτοιμοι το 2015, ούτε να έχουμε στρατηγική μετά το 2020. Thank you, And now I want to to the Minister. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον Υπουργό να απαντήσει σε αυτό το πρώτο γύρο. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Για το backloading ε, το ε, έθεσαν πολύ. Αυτό που ελπίζουμε να καταφέρουμε εμείς στην πρώτη μας είναι μια διευκρίνηση καλύτερη της οδηγίας ETS, ώστε να μπορεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει το χρονοδιάγραμμα και τις δημοπρασίες στις κατάλληλες περιόδους, ώστε να έχουμε μια καλή αγορά. Θέλουμε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση επί του φακέλου αυτού και παρότι οι προτινόμενες τροπολογίες στην οδηγία ETS ουσιαστικά είναι 21 λέξεις, φαντάζομαι ότι η όλη η διαδικασία για να επιτύχουμε συμφωνίες πρώτη ανάγνωση είναι περίπλοκη. Όλοι έχουν εκφράσει την αντίρρηση και μόνο για την έννοια του backloading. Και αυτή η τροπολογία έρχεται να διευκολύνει τα πράγματα. Κάποιες χώρες ακόμη δεν έχουν πάρει καν θέση και καλό ειδικά αυτές τις χώρες να τοποθετηθούν το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουμε να έχουμε μια κάποια βεβαιότητα γύρω από αυτή την πρόταση για να δούμε αν έχει πάρει σωστή κατεύθυνση ή όχι. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα του Ρίτσαρτ και για, για τους ρήμους του θερμοκηπίου και για κάποια άλλα ζητήματα. Έχουμε την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήρθε τον περασμένο Νοέμβρη για την αναθεώρηση νομοθεσίας του 2006, δηλαδή θα πρέπει να αυξήσουμε προσπάθειες για να μειώσουμε αυτά τα αέρια που επηρεάζουν σημαντικά το κλίμα προτείνεται μία σειρά πολιτικών λύσεων, μεταξύ άλλων να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού ή να παραταθεί, ε, μάλλον να διευρυνθούν, ε, αν θέλετε, στο πεδίο εφαρμογή ώστε να καλυφθούν οι καταψύκτες κτλ. και άλλα προϊόντα, να υπάρξουν απαγορεύσει για νέα προϊόντα και επίση απαγόρευση του HFC για οικιακούς καταψύκτες και επαγγελματικού καταψύκτες και να υπάρχουν κάποιες αλλαγές στον τρόπο ε, συντήρησης ε, των λοιπόν ε, ψυχτών. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα ανοιχτά στο τραπέζι. Πολλά είναι περίπλοκα και τεχνικά. Θα προσπαθήσουμε όμως να βοηθήσουμε κι εμείς να, ώστε να υπάρξει πρόοδο σε όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του αέρα, του ατμοσφαιρικού αέρα. Στο αστικό περιβάλλον είναι πρόβλημα αυτό. Στο άτυπο, Υπουργικό του Απριλίου θα εστιάσουμε ακριβώς στο στικό περιβάλλον. Και επίσης θα υπάρξει μια παρουσίαση για τον διαγωνισμό για τις πράσινες πόλεις που έχει διοργανώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή συζήτηση από αυτού. Για τον Τζον Λάινεν τώρα. Πολλά θέματα θέσατε. Για το Ρίο συν 20 σε διεθνές επίπεδο υπάρχει σημαντικός όγκος εργασίας, ήδη παρουσιάζει πιο πολλά και βεβαίως θέλουμε να προωθήσουμε και στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα τα πιο πολλά αποτελέσματα του στην 20. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί η ομάδα εργασίας για τα SDGs πρόσφατα επιτέλους ε, συστάθηκε και η Ιρλανδία θα κάνει ό,τι μπορεί μέσω του πρέσβη της στην ε, Νέα Υόρκη και είναι μέλος της ομάδας να προωθήσει τις θέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν θα έχουμε το Διακυβερνητικό Συμβούλιο της UNEP ε, τον επόμενο μήνα στο Ναϊρόμπι, ξέρω μένα ότι είναι μεγάλη πρόκληση, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συμφωνία για πολλά ζητήματα και χρειάζονται νέες διοικητικές δομές για τη UNEP. Πρέπει να σταθεί το υψηλό επίπεδου ε, φόρουμ των ΗΠΑ για την βιωσιμότητα ε, και είναι κάτι που απασχολεί την Προεδρία μας εξίσου. Η προτεραιότητα σε αυτή τη φάση είναι το ε, έρμο ΕΑΠ και πώς θα εφαρμοστεί. Ξέρω ότι σας απασχολεί ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα και θα ήθελα με χαρά να συνεργαστώ μαζί σας για να προωθήσουμε αυτό το φάκελο που εσείς πήγατε αρκετά μπροστά. Και για μας είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Επίσης, ε, έθεσαν διάφοροι συνάδελφοι το θέμα των κλιματικών ε, αλλαγών και τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου κατά 30%. Ναι, είναι ένα φιλόδοξο στόχο και τον συμμεριζόμεθα. Θα βάλουμε ένα σημείο στη μεσαία διατάξη του, του Υπουργικού Συμβουλίου ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν όλοι για το επίπεδο φιλοδοξίας που έχουν. Και κατά τη διάρκεια του γεύματος οι Υπουργοί Ενέργειας θα συζητήσουν μαζί με τους Υπουργούς Περιβάλλοντος το ίδιο θέμα συνεργαζόμαστε στενά με την Κομισιόν ώστε να καταλήξουμε σε μια πράσινη βίβλο για το θέμα αυτό και ελπίζουμε να είναι και η βάση της ζήτησης στο άτυπο συμβούλιο για το site της που είπε ο Chris Davis ήθιστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλά με μία φωνή η Ιρλανδία προσπαθεί όσο μπορεί να το κάνει αυτό για να ε, συμφωνεί σε μια κοινή θέση. Αυτό θα κάνουμε και εν ώψη της Μπανκόγκ. Και πιστεύω ότι ως τώρα έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο. Τώρα, σε σχέση πάλι με το ΕΑΠ, κάτι πρώτο ο Τζόου. Θα έχουμε στενή συνεργασία με όλα τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουμε και αυτό το κομμάτι που σας απασχολεί και εσάς ως μέρος του 7ου ε, ΕΑΠ. Νομίζω ότι σε όλα τα ερωτήματα. Ωραία, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο, ο Κάρθεν Φλόρενς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Προεδρεύοντα. Χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ σήμερα να μιλήσετε μαζί μας. Ε, είσαστε παλιός γνωστός ε, και χαίρομαι επίσης ε, που βρίσκεται μαζί μας η αντιπροσωπεία από την περιοχή Ρουρ. Καλώς ήρθατε. Δεν θα ήθελα κάθε μέρα να μας υποβάλλετε νέα έκθεση όπως έκανε η Κομισιόν. Θα ήθελα με περισσότερη αφοσίωση να εφαρμόσετε αυτά που αποφασίζουμε εδώ πέρα όπου και να φτάσω, ε, για παράδειγμα στην κάτω Ρινανία και στις κάτω χώρες που βρίσκονται κοντά ή ε, οπουδήποτε. Ε, πάντα αυτό με ρωτάνε και θα σας παρακαλούσα μαζί με τους συναδέλφους σας θα σας παρακαλούσα να, να κάνουμε λιγότερα αλλά καλύτερα. Για παράδειγμα, Ε, μπορεί να έχουμε νέου ανιχνευτέ καπνού, αλλά ακούμε ότι πεθαίνουν οικογένειε από μονοξίδιο του άνθρακα στο σπίτι τους ε, λόγω του, του γκριλ που χρησιμοποίησαν. Ε, επίσης ε, υπάρχει ανησυχία και τη συμμερίζομαι κι εγώ η οδηγία για τα αυτοκίνητα λόγω του ισχυρού λόμπι να αποδυναμωθεί. Έχετε περισσότερε πληροφορίε. μπορείτε να μου πείτε λίγα λόγια γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Κάρθενς Φλόρενς. Η κυρία Γκροστέτ, δύο λεπτά παρακαλώ. Alors, je ne suis pas du tout, euh, Δεν έχω συζητήσει καθόλου με τον Κάρλα Φλόρενς, με τον συνάδελφο. Όμως αυτό που ήθελα να σας πω, κύριε Υπουργέ, είναι ότι πράγματι πριν ε, καθορίσουμε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε η υπερβολητική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται και μάλιστα σωστά. Έχουμε την αίσθηση ότι ε, απλώς προχωράμε χωρίς να ανησυχούμε για το τι έχει ήδη ψηφιστεί. Για το ETS είπατε ότι χρειάζονται νέε ε, προτάσεις, είναι πολύ χαμηλή τιμή του άνθρακα και ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει μια οικονομική κρίση άνευ προηγουμένου. Εμένα με απασχολεί ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα γιατί η ο κλάδος της βιομηχανίας, οι επιχειρήσεις ε, χρειάζονται μια νομική ασφάλεια και η μεγαλύτερη ανησυχία του είναι ότι συνεχώ ε, το κοινοβούλιο μα ε, αμφισβητεί τα όσα έχουν ψηφιστεί. Και θέλει πάντα να προχωρά χωρίς να ξέρει αν τηρούνται ε, τα προηγούμενα, όσα έχουν ήδη ψηφιστεί. Αυτά είναι τα ζητήματα που θέλω να θέσω και εφόσον μιλάμε και για το ETS, βεβαίως και όλο και περισσότερο τα κράτη-μέλη προσφεύγουν στον άνθρακα. Λαμβάνοντα υπόψη και τα όσα έχουμε πει για τι εκπομπέ του διευθυντή του άνθρακα, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Υπουργέ, αν ε, προτίθεστε να ασχοληθείτε με αυτό το μεγάλο και ιδιαίτερα πολύπλοκο και λεπτό ζήτημα τη ε, της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Υπουργέ, για αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το σύστημα εμπορίας εκπομπών ε, και τις αερομεταφορές. Ε, η δουλειά δεν θα πρέπει να γίνει εντός της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας. Φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ. Ξέρω ότι παραδοσιακά η Ιρλανδία έχει πολύ καλές σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αδερφικές σας σχέσεις με, το Ηνωμένο με, με τις Ηνωμένε Πολιτείε, ώστε να καταλήξετε σε μια καλή συμφωνία. Και επίσης ε, όταν ε, μιλήσετε με τον Λευκό Οίκο μήπω μπορείτε να του αναφέρετε και τη διάσκεψη site ε, στην Bangkok διότι κατά την τελευταία διάσκεψη υπήρχαν κάποιε παρανοήσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή και την Αμερικανική Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία. Ε, άλλωστε όμως έχουμε τους ίδιους στόχους. Η δεύτερη με έχει να κάνει με την κοινή γεωργική πολιτική. Ε, ενώ όσο μιλάμε, η Επιτροπή Γεωργίας έχει αποδυναμώσει τις περισσότερες ε, προτάσεις ε, περί πρασινίσματος, περί περιβαλλοντικής διάστασης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φοβάμαι ότι και οι Υπουργοί Γεωργίας θα κάνουν το ίδιο. η ερώτηση προς εσάς είναι, θα παρέμβει το Συμβούλιο Περιβάλλοντος πάνω στη κοινή γεωργική πολιτική, διότι αν δεν το κάνει αυτό δεν θα πετύχουμε ποτέ τους ε, στόχους ε, για το κλίμα και τη βιοπικιλότητα που έχουμε θέσει, ε, για τους οποίους είναι υπεύθυνο και το Συμβούλιο. Τρίτον, περιμένουμε μια στρατηγική περιπλαστικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιθανή απαγόρευση ή ε, τέλη για τις ε, πλαστικές σακούλες ε, ελπίζω να συμπεριλαμβάνονται. Ξέρω ότι οι έχουν... Η Ιρλανδία έχει πάρα πολύ καλές εμπειρίε. Μήπω μπορείτε να μας μιλήσετε για τις εμπειρίε σας και τι θα προσπαθήσετε να πετύχετε εντός του Συμβουλίου. Τέλος, όσον αφορά τους στόχους βιώσιμη ανάπτυξη σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, φαίνεται να υπάρχει πάντα μια σύγκρουση ανάμεσα σε αυτού που ασχολούνται με την ανάπτυξη και σε αυτού που ασχολούνται με το περιβάλλον. Μπορείτε να μα το αναπτύξετε αυτό. Ευχαριστώ, Καλ Σλίτερ. Ε, ευχαριστώ, καλώ ήρθατε. Ε, όπως ε, αναφέραμε και πριν, υπάρχει το θέμα της ανακύκλωση των πλοίων, ε, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ και στα ελαφριά εμπορικά αυτοκίνητα, τα LCV εάν καταφέρετε κάτι, αυτό θα είναι καλό για τις επιχειρήσεις, θα είναι καλό για το περιβάλλον, θα είναι καλό και για ε, τους καταναλωτές ε, κάθε ε, λογαριασμός ε, ε, ηλεκτρολόγου ή υδραυλικού στην Ευρώπη θα είναι χαμηλότερος εάν αν μπορείτε να κάνετε μια τολμηρή πρόταση πάνω στα ε, ε, LCV και δεν ε, θέλουμε απλά να επικεντρωθούμε στους παλιωμοδίτες παραγωγές παραγωγούς ε, που δεν ξέρουν τίποτα περί ε, εξαγωγών. Ελπίζω να μπορέσετε να βρείτε ε, θετική πλειοψηφία ώστε να μπορέσετε να έχετε μια φιλόδοξη πρόταση. Τέλος, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα, την προετοιμασία της συνάντησης στην Πολωνία κλπ. Παλαιότερα είχαμε την τάση όταν έρχονται οι Ευρωπαίοι Υπουργοί στις ε, διεθνείς αυτές συναντήσεις ε, συνομιλούν πολλή ώρα μεταξύ τους ε, για να βρουν λύσεις και ομοφόνες αποφάσεις. Ελπίζω ε, να, έχετε, να προγραμματίσετε να συνομιλήσουν οι υπουργοί και με υπουργού εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε και του άλλου. Ε, δεν ξέρω πώ μπορεί να γίνει αυτό, αλλά αν, μπορέσετε, αν βρείτε έναν τρόπο αυτό θα μπορέσει να επηρεάσει τι ε, παγκόσμιε πολιτικέ για την αλλαγή του κλίματο. Αυτό ζητώ από εσά. Ευχαριστώ πολύ. Κορίν Λεπά, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μα. Ε, δύο ζητήματα. Πρώτον, τι θα γίνει με το κείμενο που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση για τους ε, ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, εφόσον η Επιτροπή αποφάσισε να ξεκινήσει από την αρχή όλη τη διαδικασία, αν κατάλαβα καλά από αυτή την περίπλοκη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε χθε. Τι σημαίνει λοιπόν με αυτό. Δεύτερον, σκοπεύετε να επηρεάσετε την Επιτροπή για την λήψη μέτρων για ορισμένα προϊόντα των οποίων ε, έχει αναγνωριστεί πλέον η τοξικότητα. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες ουσίες που επηρεάζουν τις ε, Ευχαριστώ και η Κρίστα Κλάς ε, δυστυχώς δεν την είδα πριν. Θα ήθελα λοιπόν να τη ζητήσω συγγνώμη. Καλά, ναι, δεν δε φαίνομαι από εδώ νομίζω. Ε, κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε πολύ σύντομα στο ζήτημα ILOC και ε, σημειώνω ότι οργανώνεται δικό σας ε, σεμινάριο τον ε, Ιούνιο ε, και θέλετε να παραδώσετε το θέμα μετά και στην Λιθουανική Προεδρία. Ε, δημιουργούμε νέους ε, παράγοντες ε, στον τομέα του και Είναι θεωρητικό αυτό, χρειαζόμαστε αντικειμενικά κριτήρια. Πρέπει δηλαδή να έχουμε και την υποστήριξη της έρευνας. Ε, ε, μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά ξαφνικά με την πρόταση της Κομισιόν ε, μειώνουμε τις φιλοδοξίες μας ε, και συμβαίνει αυτό που είπαν ο Καλχάνης Φλόρενς και η Φρανσουάς Κροστέτ, ότι χρειαζόμαστε αξιοπιστία στην πολιτική και σε αντίθεση με τον ε, συναδελφό Μπράντι θα ήθελα να πω ότι η συμβατότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής με τη γεωργική πολιτική δεν ε, υπάρχει ακριβώς, διότι ε, στη γεωργική πολιτική μιλάμε για ε, περιοχές, για εκτάσεις περιβαλλοντικής εστίασης, ενώ από την άλλη μιλάμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος άλλα θέματα τα οποία δεν ταιριάζουν με αυτά Παρακαλώ να το έχετε υπόψη σας αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κλάς. Ε, πολύ ευχαρίστω σας κοιτώ πάντα. Ε, ωραία τώρα κοιτώ από ε, την άλλη μεριά η Μαργαρέτα Ούλσκοκ. Ε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ που είσαστε παρόν κύριε Υπουργέ. Έχουμε θέσει πολλές ερωτήσεις ε, και έτσι έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν τον κατάλογο, αλλά θα ήθελα να επαναλάβω. Επαναλαμβάνω, ευχαριστώ ε, κύριε Υπουργέ που είσαστε παρόν. Ε, σε αυτό το στάδιο της συζήτησης επαναλαμβάνει κανείς ερωτήσεις, διότι νομίζω ότι τα ίδια θέματα ενδιαφέρουν πολλούς από τους ε, συναδέρφους ε, εδώ. Ε, θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβω κάποια ερωτήματα που τέθηκαν. Σε όλες τις πολιτικές ομάδες συζητάμε αυτή τη στιγμή το σύστημα εμπορίας εκπομπών και ξέρουμε ότι το πολυσυστημένο αυτό σύστημα το οποίο είναι σημαντικό μέρος της συμφωνίας του Κιώτο που όμως δεν εφαρμόζουν πολλές χώρες αλλά που ξεκινούν να εφαρμόζουν νέα κράτη όπως είναι η Αυστραλία, η Κίνα, η Νότια Κορέα, η Καλιφόρνια κλπ. Τώρα λοιπόν που επεκτείνεται το σύστημα αυτό, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε έναν καλό συμβασμό σχετικά με το backloading όπως ε, και άλλοι ευρωβουλευτές, θα ήθελα να ακούσω πώς βλέπετε εσείς τη δυνατότητα να υπάρξει υποστήριξη για το backloading, ώστε να μπορέσουμε αργότερα να έχουμε μία μακροπρόθεσμη πρόταση σχετικά με το πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να περιορίζουμε τις εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Ένα σχετικό φόρο θα ήταν πολύ καλό πράγμα, αλλά θα ήταν πολύ δύσκολο να περάσει στο Συμβούλιο. Η άλλη μου ερώτηση έχει να κάνει με τις ε, εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα από τα οχήματα. Ε, ξέρουμε ότι οι υπολογισμοί που έγιναν σχετικά με τις εκπομπές, το κόστος Ξέρουμε ότι οι υποθέσεις που είχαν γίνει τότε σχετικά με τα νούμερα έχουν αλλάξει πολύ έκτοτε. Υπάρχει μάλιστα υποψία ότι ο σχετικός κλάδος δεν ανέφερε, δεν χρησιμοποίησε τα, τα σωστά στοιχεία. Ε, τώρα λοιπόν λέγεται ότι δεν θα πρέπει να γίνουμε πιο φιλόδοξοι, απλά να ε, κάνουμε κάποιες ε, μικρές ε, προσαρμογές. Ε, θα πρέπει δηλαδή να διατηρήσουμε τις πολύ γενναιόδορες πιστώσεις που είχαμε τότε. Και αυτό σε μια εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει κρίση. Τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε πιο φιλόδοξα σχέδια όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον Υπουργό για την παρουσία του. Δύο ερωτήσεις συγκεκριμένα θα ήθελα να θέσω. Η πρώτη αφορά τις όλες τις ρυθμίσεις για, τις, ε, για του θερμοκηπίου και σε αντίθεση με αυτά που είπε ο κύριος Ρούσκοφ. Η δική μου άποψη διαφέρει, θα έλεγα, σχετικά με την ερμηνεία του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Δεν πιστεύω ότι έχουν γίνει ουσιαστικές, ουσιαστικά βήματα μπροστά με τις δηλώσεις στον Παλί και την ανάληψη α, κοινής ευθύνης, κοινής μεν διαφοροποιημένης δε. Common but differentiated responsibility. Αυτό όμως σημαίνει δεν υπάρχει απόλυτη ισότητα, ε, ισονομία και δικαιοσύνη. Εν προκειμένου πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Να αλλάξει η δομή του ETS ώστε να λάβουμε υπόψη και την ανάγκη για δικαιοσύνη και ισότητα. Δεύτερο ερώτημα. αντιμετωπίζουμε τη θέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή που ήδη έχει λάβει πολύ σημαντικά καταστρεπτικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να σπαταλήσουμε πλέον ούτε ένα δευτερόλεπτο. Θα πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση, ε, μια επίγουσα κατάσταση και πολύ βλαπτική κατάσταση. Εκπλήσωμε όταν βλέπω ότι η κοινή αγροτική πολιτική δεν αναφέρεται καν σε αυτό το ζήτημα. Ενώ είναι υπερεπίγον να υπάρξει ισχυρό συντονισμό για την επίλυση αυτού του προβλήματο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε έτσι τον κύκλο των ερωτήσεων. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, συνεισφορές σας και για τα ζητήματα που εγκουθήξατε, που είναι εξαιρετικά σημαντικά. Νομίζω ότι Κάποιο είπε ότι του πέσαν τα μαλλιά με τα όσα έχει ακούσει. Εγώ νομίζω ότι μόνο εγώ το έχω αυτό το πρόβλημα. Ελπίζω να μην το έχετε κι εσεί. Σε ό,τι αφορά τώρα την εφαρμογή, είναι κρίσιμη σημασία σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συμφωνώ λοιπόν με τα όσα είπατε, η κυρία Ροζέτα αυτό είπε. Και ε, δίνουμε και μεγάλη έμφαση σε αυτό το τομέα στο πλαίσιο του 7ου EAP. Στην Ιρλανδία δυσκολευθήκαμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα, αλλά και να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες δομές για την αυστηρή εφαρμογή του περιβαλλοντικού νομοθετικού πλαισίου και καταβάλουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες για να ευθυγραμμιστούμε. Ε, χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι πολλά κράτη-μέλη της δεν θα ε, συμμορφώνονταν με τις ε, διεθνείς κατάλληλες πρακτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας βοηθάει λοιπόν ε, να το κάνουμε αυτό. Είναι κάτι που το αναγνωρίζουμε όλοι και είναι προφανές. Σας Παροτρύνω λοιπόν να συμβάλλετε κι εσείς ε, στην ε, υλοποίηση του 7ου EAP εφόσον και ένας από τους κρίσιμους τομείς είναι η υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής της υφιστάμενης ε, περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Και ελπίζω να συνεργαστούμε στενά για αυτά τα ζητήματα. Για το ETS, από γενικής πλευράς νομίζω ότι πράγματι είναι ένα τεχνικό ζήτημα το κοινοβούλιο είναι αυτό που θα αποφασίσει αν ε, θέλει το ETS ε ή όχι. Και ελήψη αυτού πρέπει να προτείνει κάποιο άλλο σύστημα. Αυτό είναι ο δικό σα ρόλο και είναι και μεγάλη πρόκληση βεβαίω. Για να βρούμε μια εναλλακτική λύση ως προς το υφιστάμενο σύστημα. Αυτό θα γίνει βέβαια μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ο καλός μου φίλος κ. Γεμπράντη, ανέφερε ότι υπάρχει πράγματι μια στενή συνεργασία και δεσμοί με τις ΗΠΑ. Ε, πάνω από 40 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες δηλώνουν ότι είναι Ιρλανδοί, επομένως είναι σίγουρα και αυτό σε ένα σημαντικό θεσμό και σίγουρα θα έχουμε μια επίσκεψη μάλλον διήμερη στη ΣΥΠΑ, εφόσον προεδρεύουμε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να βελτιώσουμε και τις ε, σχέσεις μας. Αλλά σίγουρα σε ό,τι αφορά το θεματολόγιο για την κλιματική αλλαγή θα ε, ε, θα δούμε αν ε, κατά πόσο ο κύριος Ομπάμα ενδιαφέρεται για τέτοια ζητήματα κλιματικής αλλαγής και αν ενδιαφέρεται να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με την προηγούμενη του θητεία. Ίσως μπορεί να τα πάει καλύτερα και με το Κογκρέσο. Αναφερθήκατε σε διάφορα μέτρα που έχει υλοποιήσει η Ιρλανδία που ήταν και επιτυχή μάλιστα. Εδώ και μια δεκαετία το έχουμε κάνει αυτό. Πώς δηλαδή μπορεί να ένας, ένα αντίτιμο, ένας φόρος, ένα τέτοιο μέσο να έχει μεγάλη ε, επίδραση στη συμπεριφορά του καταναλωτή, αλλά και ως προς ε, την ε, αποδοτικότητα των πόρων σε σχέση με τις πλαστικές σακούλες. άλλα ζητήματα που αναφέρθηκαν ε, στο greening, στην ε, γεωργική πολιτική. Ε, υπάρχει ευρεία συνένεση για το greening στον πρώτο πυλώνα με τα τρία κριτήρια. Όμως υπάρχουν και πολλά ανοιχτά ζητήματα για την ενεργοποίηση, τα ποσοστά και την ευελιξία που θα δοθεί στα κράτη-μέλη. Βεβαίως και τα κράτη-μέλη επιθυμούν την ευελιξία σε ορισμένες περιπτώσεις βάσει των τοπογραφικών χαρακτηριστικών και του γεωγραφικού πλαισίου. Αυτά τα θέματα είναι γνωστά στην Ιρλανδική Προεδρία. Και σίγουρα και εγώ είμαι στην επαφή με τον κύριο Κόβλνε, Υπουργό Γεωργία και πρώην Ευρωβουλευτή, ε, που είναι βεβαίω ο πλέον ειδικό στου ζητήματα γεωργία. σίγουρα και ο ίδιος αναγνωρίζει τη σημασία της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα δω τι πρόοδο θα σημειώσει εκείνος και τι πρόοδο θα μπορούμε να σημειώσουμε μαζί για συμβιβασμού ε, που θα αποδεχόμαστε όλες. Γιατί η κυρία Λαπάζ αναφέρθηκε στο θέμα των γενετικώ τροποποιημένων οργανισμών. Αναγνωρίζουμε την ε, σημαντική πρόοδο που σημαίνει η Ιδανική Προεδρία. Είναι δύσκολη η συμφωνία αυτή. Έχουμε εξετάσει τις προτεραιότητές μας ε, για την Προεδρία και δεν βρήκαμε πολλά ενδείξεις ε, προόδου και συμφωνίας, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε. Έχουμε 126 ζητήματα που έχουμε ε, προσδιορίσει. Θα δούμε σε ποια μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. ο Κρις Λεκλάς το Έχουμε εννέα ομάδες εργασίας που, έχουμε, που έχουν προγραμματιστεί και μια συζήτηση προσανατολισμού στο Συμβούλιο για αυτό το φάκελο. Ελπίζουμε λοιπόν να υπάρξει κάποια πρόοδο και εδώ. Αγαπητέ Οσμπροκ, ξεκινήσαμε συζήτηση στο Συμβούλιο με την Ελβετία για το ETS. Και θα έχουμε και μια παρόμοια πρόταση με την, για την Αυστραλία στην ομάδα εργασία την Παρασκευή και αυτές οι συνδέσεις μπορούν μόνο να ενισχύσουν το ETS. Ο καλός μου φίλος Κάρις Λούιζερ ανέφερε το επίπεδο φιλοδοξίας μας ό,τι αφορά τα ελαφρά οχήματα και τα φορτηγά. Ε, και εσείς ε, βεβαίως ε, έχετε την ευκαιρία να πείσετε τους συναδέλφους σας για το επίπεδο φιλοδοξίας και σας εύχομαι καλή τύχη. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει ένα συμβιβασμό και από τις δύο πλευρές. Όμω. οι εισηγητέ και συνεισηγητέ εδώ καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες και βεβαίω το επίπεδο φιλοδοξίας είναι κάτι υποκειμενικό. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε γιατί ε, και ο κλάδος ε, αυτός ε, χρειάζεται την ασφάλεια και τη βεβαιότητα καθώς και το περιβάλλον. Για όλους αυτούς του τομείς λοιπόν είναι καλύτερο να υπάρξει συμφωνία παρά να μην υπάρξει. Συμφωνώ μαζί σας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν πάντα, δεν είναι πάντα, δεν έχει πάντα ενιαία θέση ε, στις διεθνείς συνδιασκέψεις. Ούτε στην Τόχα κρατήσαμε την πιο ενιαία μας στάση μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτό βέβαια δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, ωστόσο μαθαίνουμε από αυτές τις εμπειρίες και ελπίζουμε στις μελλοντικές συνδιασκέψεις στις οποίες θα συμμετάσχουμε να μην ισχύσει κάτι τέτοιο. Αυτό θα πρέπει να γίνει στο μέλλον, να είμαστε όσο δυνατόν πιο ενιαίοι ή να έχουμε μια συμπεφωνημένη στάση, αν όχι ενιαία. Ο κύριος Πρόντι. Μεγαλύτερη φιλοδοξία είπατε ότι χρειάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καινοτομία και την κλιματική αλλαγή. Εγώ προσπαθώ να διευκολύνω αυτές τις συζητήσεις ε, ως ε, αμερόληπτος ε, συμμετέχων σε αυτές τις διαδικασίες. Θα δούμε και τι θα γίνει στην άτυπη συνεδρίαση του Απριλίου Ελπίζω να μας βοηθήσει αυτό να κατανοήσουμε τη στάση ε, των επιμέρους κρατών μελών και που θέτουν τον πύχη της φιλοδοξίας για το μέλλον. Σίγουρα έχετε δίκιο για τα όσα πρέπει να επιτύχουμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο πλαίσιο των μελλοντικών διεθνών πραγματεύσεων είμαστε υπεύθυνοι και εμεί, ευθυνόμαστε μάλλον για το 12-13% των ε, εκπομπών ε, αερίου του θερμοκηπίου. Εμεί είμαστε οι καλοί. Βεβαίω και θέλουμε να ενθαρρύνουμε του υπολείπου ε, και να φτάσουμε το 2015 που είναι μια σημαντική πρόκληση, παρόλο που έχουμε ηγετικό ρόλο, ίσως θα πρέπει να το κάνουμε ακόμα παραπάνω. Και αν θέλουμε να φέρουμε με το μέρος μας τους υπόλοιπους φορείς και παίκτες μέχρι το 2015, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Είναι μεγάλη πρόκληση. Και παρόλα αυτά να, να διατηρήσουμε και μια ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα της κοινή αλλά διαφοροποιημένης ευθύνη για τις διεθνείς συζητήσεις και οι 195 θα συνυπογράψουν το 2015. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόκληση λοιπόν. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για το επίπεδο φιλοδοξία μας, αλλά όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στη Δόχα, Εάν θέλει κάποιος ε, να, να συγκαλέσει τους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων το 2014 ενώ του 2015 είναι και αυτό ένα σημαντικό βήμα. Και θα το τονίσει αυτό και όταν θα συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ τον Μάρτιο. Η αλλαγή στην οτροπία, στη συμπεριφορά που αναφέρθηκε προηγουμένως, εμείς στην Ιρλανδία με αυτό τον ε, φόρο ή το αντίτιμο για τις πλαστικές ε, σακούλες, ε, για το σύστημα φορολόγησης του νερού με έναν πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, έχει αλλάξει τη, τη συμπεριφορά των πολιτών. Το 80% των πωλήσεων αυτοκινήτων το 2012 και 2011 δείχνουν ότι πλέον οι καταναλωτές στρέφονται προς τα οχήματα με μικρότερες εκπομπές. Λόγω και της αλλαγής ε, στο φορολογικό σύστημα. Έχει δώσει λοιπόν κίνητρο ε, στους πολίτες να κάνουν το σωστό για το περιβάλλον και να αγοράσουν και ένα αυτοκίνητο καλής ποιότητας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι λοιπόν που μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να μάθουμε ο ένας από τον άλλον. ελπίζουμε με όλους αυτούς τους τρόπους να αυξηθεί και το επίπεδο φιλοδοξίας. Είτε αυτό γίνει με τα οχήματα για τα φορτηγά, είτε ε, με τις ουσίες στο νερό. Αυτό θέλουμε να επιτύχουμε, να αυξήσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας. Ευχαριστώ. Herr Minister, vielen Dank für die... Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ <clears throat> για τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις μας να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο για τις εργασίες σας στο επόμενο εξάμεινο. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι έχετε πολλή δουλειά. Υπάρχουν πολλά θέματα επιτάπητος και μάλιστα αποφασιστική σημασία θέματα με τα οποία θα υπολογιστεί η αξιοπιστία μας και εν μέρει όσον αφορά ε, τουλάχιστον ε, το σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών θα φανεί και η καλή λειτουργία της Ευρώπης. Όλοι λοιπόν φέρουμε σημαντική ευθύνη και εσείς στο Συμβούλιο και εμείς στο Κοινοβούλιο. Είμαι βέβαιος όμως ότι τα πράγματα θα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι θα επισκευάσουμε αυτά που χρειάζονται επισκευή και θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τα άλλα. Ο συνάδελφος Καρλ Χάινς Φλόρενς αναφέρθηκε ε, στο θέμα της στήρησης ε, και της εφαρμογής της νομοθεσίας. Ε, θα... Είχαμε ε, προσκαλέσει εδώ και τον ε, ε, ειδικό πρόσωπο για την κατάρριξη τη γραφειοκρατίας, τον κύριο Στόιμπερ και έχουμε υπόψη μα και όλα αυτά που είχαμε συζητήσει τότε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα βρείτε πάντα μια ανοιχτή πόρτα. Είσαστε πάντα ευπρόσδεκτος. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι ολοκληρώσαμε και τη σημερινή συνεδρίαση. Θα τα πούμε αύριο στις 10. Θα συνεχίσουμε με το backloading και οι συντονιστές ε, θα ξεκινήσουν στις 9. Καλό βράδυ.